Αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε τις εργασίες μας για σήμερα το απόγευμα και πάλι. Και στην ημερήσια μας διάταξη έχουμε δύο πολύ σημαντικές ακροάσεις ε, σε μια αίθουσα που δυστυχώς δεν είναι κατάλληλη ούτε για ψηφοφορίες ε, ούτε για τόσο σημαντικές ακροάσεις. Γι' αυτό και θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τους συναδέλφους οι οποίοι δεν βρίσκουν θέση να καθίσουν, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, όσοι όμως θέλουν να παρακολουθήσουν τις εργασίες μας και έτσι εκτάκτο, εκτάκτο. Ε, αν είστε όρθιοι και δεν έχετε ένα κάθισμα, τότε εντάξει, σας δίνουμε την άδεια να πάρετε τις θέσεις, να καταλάβετε τις θέσεις των απτυρωματικών μελών με πράσινες ε, καρτελίτσες, έτσι. Λοιπόν, τελειώσαμε το τεχνική σε αυτής φύσεως σημείο που είναι όμως σημαντικό. Η Επιτροπή που μας ε, που έχουμε την εισήγηση για την απόσπαση των εργαζομένων Σήμερα το πρωί οργάνωσε ήδη μια ακρόαση για το ίδιο θέμα. Αυτό Μάλλον τώρα ενημερώμενοι γι' αυτό και δυστυχώς ε, δεν φαίνεται να λειτουργεί καλά επικοινωνία ανάμεσα <laughs> μας. Και θα τα πω αυτά στη διάσκεψη των Προέδρων. Ο κ. Κρίστανσεν ενώ μεταξύ μου ζήτησε κάτι. Επειδή έχει μια ομάδα από διαφωνικό σταθμό που τον, τον ακολουθεί για να ε, μαγνητοφωνήσει τις ε, συζητήσεις και λέει ακριβώς μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όχι όμως δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα γι' αυτό αν έχετε ζωντανή αναμετάδοση στο δανέζικο ραδιόφωνο να μην εκπλαγείτε. Αυτά λοιπόν και έχουμε και τα συνδικάτα των εργαζομένων έχουμε τα σχετικά κείμενα δόθηκαν σε εσά, σας, στα μέλη και Ζητούν και οι υπόλοιποι να έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Εντάξει, δεχτήκαμε και έχουμε αρκετούς εμπειρογνώμονες μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Σύντομα, σύντομα, το λόγο θα λάβει η συγκήτριά μας, ε, κυρία Δανούτα Ζασλόβιασκα, για να μας κάνει μια εισήγηση, αρχική τοποθέτηση και δέκα λεπτά μετά για να απαντήσουμε στα συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία και έχουν τεθεί. Η κυρία Ζασλόβισκα έχει το λόγο. Πριν να έρθουμε τώρα στην οδηγία, θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένες πτυχές και οργανωτικές πτυχές και αναφερθήκε η Πρόεδρος στη σημασία αυτών και χρειάζεται όλοι να έχουν πρόσβαση να μπορούν να ενημερωθούν για τη συνάντησή μας. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να συμμετάσχουμε στη συνάντηση της ΣΥΜΚΟ γιατί ψηφίζαμε. Λυπάμαι πάντως διότι η Επιτροπή μας δεν ε, μας ενημέρωσε για αυτή την ακρόαση αντίθετα με εκείνο που έκανε η ΙΜΚΟ δηλαδή και δεν ασχοληθήκαμε όπως πρέπει και δίκαια με όλους τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι κανονικά θα ήθελαν, θα έπρεπε να συμμετάσχουν στη συνάντηση αυτή και λυπάμαι πάρα πολύ για ό,τι συνέβη. Να έρθουμε τώρα στις τεχνικές πτυχές της οδηγίας. Κυρίες και κύριοι, η 96 κάτω 71 οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων προκαλεί πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα μπορούμε και συμμετέχουμε σε μια ακρόαση στην οποία συμμετέχουν επίσης εμπειρογνώμονες στον τομέα αυτό. Η οδηγία στον τομέα εφαρμογής της πρέπει να είναι αποτελεσματική και αυτό επαναλαμβάνω για την απόσπαση των εργαζομένων στο πλαίσιο επιρροχής επισιών. Έχουμε δύο στόχους ε, της οδηγίας. Η πρόθεση είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε όσοι προσφέρουν υπηρεσίες να μπορούν να το κάνουν ε, κατά από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ε, και να γίνουν σεβαστά και όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Οργανώθηκαν πολλές ε, συναντήσεις με εκπροσώπους του κλάδου αλλά και εργοδότες ε, και μας είπαν μάλλον καταλάβαμε ότι τα προβλήματα που έχουν σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας είναι πολυάριθμα. Πάνω απ' όλα για την εφαρμογή και πώς κανείς μπορεί να έχει αυτές τις συνθήκες κατάλληλες εργασίες ε, την αξιοπιστία των επιχειρήσεων. Ε, ορισμένους που απλά και μόνο δανείζουν την ετικέτα τους, το όνομά τους ε, και την ε, δίθεν πρόσληψη. Εδώ λοιπόν όλες οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αποτελούν όλες, επαναλαμβάνω, καλή λύση, άριστη λύση για να λυθεί το πρόβλημα της απόσπασης των εργαζομένων. Και δεν γνωρίζω αν αυτές οι ρυθμίσεις, οι διατάξεις είναι αρκετά διάφανες. Ένα μεγάλο μέρος των αμφιβολιών μου ε, της απίφθηνας του συμμετέχοντες στην ακρόαση εδώ σήμερα. Θα ήθελα να συντάξουμε ένα κείμενο σαφές, διάφανο με όλες αυτές τις διατάξεις, τις ρυθμίσεις και ελπίζω ότι θα βοηθήσουμε με τη σημερινή μας απογευματινή συνάντηση για να διαλύσουμε κάθε αμφιβολία όσο τη δυνατότητα καλής τεχνικής λειτουργίας αυτής της οδηγίας από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ. Εδώ ολοκληρώνω ώστε να μπορέσουν οι να λάβουν το λόγο. Ναι, και τώρα με τη σειρά που έχω εδώ μπροστά μου θα δώσουμε το λόγο στους τέσσερις ε, προσκεκλημένους μας. Κύριε Συγήτρια, να σας υπενθυμίσω ότι αυτό γίνεται τώρα κάπως σε διαφορετικό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποσύρει το κείμενο που παράλληλα με το δικό σας είχε ε, ε, δώσει το Μοντιδίο και έτσι θα πρέπει να δούμε σήμερα τη δική σας την έκθεση και το λόγο έχει ο κύριος Βέρνερ Μπίλεν. Είναι πολιτικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζομένων στην Σικοδομές και την Ξυλία. Έχει το λόγο ο κύριος Μπίλεν για 10 λεπτά περίπου. Ευχαριστώ. Εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Εργαζομένων ε, στις οικοδομές και το τομέα της ξυλίας. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για την πρωτοβουλία αυτή. Είναι πολύ σημαντικό ε, να ανταλλάσσουμε προφορίες με τους εμπλεκόμενους φορείς και είμαστε ρητεθειμένοι να υπάρξουν ε, και δημιουργικές λύσεις και να συμφωνήσουμε σε συμβιβασμού. Λόγω του περισμένου χρόνου ομιλίας έχουμε υποβάλει τις απαντήσεις στις ερωτήσεις μας ε, γραπτά. Τα έχουμε στείλει στη γραμματεία της Επιτροπής, της Επιτροπής σας. Υποθέτω ότι η γραμματεία θα σας δώσει, θα σας έχει ήδη διανύμει τις γραπτές μας αντιδράσεις. Οπότε μπορείτε, αν θέλετε, να κάνετε περαιτέρω ερωτήσεις, να μας στείλετε ένα email και θα στείλουμε γραπτές απαντήσεις. Πριν ξεκινήσω, να πω ότι παρά το ότι χαιρόμαστε που έχει προσκληθεί ο τομέας των κατασκευών, αλλά δεν είναι μόνο δικό μας θέμα. Πολλοί από τους συναδελφούς μας σε άλλους τομείς, ε, στα σφαγεία και σε άλλους τομείς αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Γι' αυτό σήμερα δεν θα μιλήσω από πλευράς ε, του οργανισμού μου, αλλά από πλευράς όλων των συνδικάτων. Δηλαδή ε, όλα όσα καλύπτει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων. Αν εξετάσετε τις ερωτήσεις, θα ήθελα να συγκεντρώσω την προσοχή μας στις πιο σημαντικές. ερώτηση 2, για παράδειγμα. Θέτει το ερώτημα, ποιο είναι το ουσιαστικό θέμα πριν ε, επιλύσουμε το πρόβλημα πρέπει να το ορίσουμε. Δηλαδή το πρόβλημα καταστρατήγησης. Είναι πολύ μεγάλος ο κατάλογος, ε, μην εκπλαγείτε λοιπόν. Πολλοί εργαζόμενοι όταν αποσπώνται σε άλλη χώρα δεν έχουν την παραμικρή ιδέα για τους όρους απασχόλησής τους και τις συνθήκες. Έχουν κάποιες αόριστες ε, αντιλήψεις τι περίπου θα μπορούσε να λάβουν ως αποδοχές αλλά γενικώ δεν έχουν την παραμικρή ιδέα τι κανονισμοί ισχύουν στις χώρες υποδοχή. Σοβαρή έλλειψη λοιπόν ενημέρωση. Αυτό είναι λοιπόν το βασικό θέμα της οδηγίας για την απόσπαση που λέει σαφώς ότι τα κράτη-μέλη έχουν την υποχρέωση να παράσχουν πληροφόρηση. Πολύ συχνά υπάρχει αυτή η ενημέρωση, ας πούμε σε κάποιο κρυμμένο ιστοτόπο, σε μια γλώσσα που δεν την γνωρίζουν, όπου κανένας ε, οικοδόμος δεν πρόκειται να πάει. Υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες από τη βάση, είτε από κοινωνικούς εταίρους, μέσω του κοινωνικού ταμείου, μέσω άλλων οργανισμών. Έτσι υπάρχουν κάποια site, κάποια φυλάδια, λειτουργούν αρκετά καλά. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι αποσπασμένοι δύσκολα έχουν πρόσβαση και τα συνδικάτα έχουν τα δικά τους φυλάδια. Ο πιο αποτελεσματικός λοιπόν τρόπος ε, ενημέρωσης δεν είναι μέσω των κρατών μελών, δυστυχώς μέσω των κοινωνικών εταίρων γίνεται αυτή η ενημέρωση παρόλο που δεν είναι ευθύνη μας. Δεύτερο πρόβλημα. Θεωρητικά, σύμφωνα με την οδηγία 91-534, 533 ο εργοδότης πρέπει να δώσει σαφή ενημέρωση για το ποιοι οι κανόνες, ποιες συνθήκες πρέπει να ισχύουν και τι δικαιώματα έχει ο εργαζόμενος. Πρέπει να αναφέρονται στο συμβόλαιο. Το πρόβλημα με την οδηγία αυτή και είναι οδηγία που έχουμε πολλά χρόνια τώρα. Η οδηγία αυτή δεν εφαρμόζεται καθόλου. Είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό. Μια οδηγία λοιπόν που στην ουσία είναι νεκρό γράμμα. Βεβαίω προβλέπει σημαντικέ υποχρεώσει για του εργοδότες, για ενημέρωση. Αλλά δεν εφαρμόζεται. Οι περισσότεροι λοιπόν αποσπόμενοι φεύγουν από τη χώρα προέλευση χωρίς ενημέρωση. Όταν αποσπαστούν στο εξωτερικό είναι πολύ απομονωμένοι, υπάρχει πολλή πίεση. Δεν είναι λοιπόν σε θέση να διαμαρτυρηθούν γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι αν διαμαρτυρηθούν είτε θα τους επιβληθούν πρόστιμα, άλλες κυρώσεις ή θα τους στείλουν πίσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα των αποσπασμένων όταν διαμαρτύρονται. Ή ο εργοδότης εξαφανίζεται. Ζουν λοιπόν πολύ απομονωμένοι. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι δεν γνωρίζουν τη γλώσσα, τον πολιτισμό της χώρας ε, υποδοχής. Δεν ξέρουν πού πρέπει να στραφούν σε περίπτωση διαμαρτυριών, δεν ξέρουν ότι υπάρχουν επιθεωρητές εργασίες, δεν ξέρουν ποιος είναι ο ρόλος των ε, συνδικάτων στη χώρα αυτή. Τα συνδικάτα λοιπόν πρέπει να τους ψάξουν τους αποσπασμένους. Οι επιθεωρητές πρέπει να τους ψάξουν. Οι αποσπασμένοι δεν πάνε μόνοι τους σε ένα συνδικάτο. Από ό,τι έχουμε δει έρχονται σε εμά μόνο εάν δεν έχουν πληρωθεί για τουλάχιστον τρει μήνες, για έξι μήνες. Οπότε ζουν σε απάνθρωπες, απάνθρωπες συνθήκες. Οπότε προφανώς αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης έχει εξαφανιστεί. Ο έλεγχος επίσης είναι σοβαρό πρόβλημα. Ήδη στη χώρα προέλευσης δεν γίνεται τίποτα. Δεν υπάρχει σύστημα ενημέρωσης, δεν υπάρχει διαρθρωμένη ανταλλαγή πληροφοριών, οπότε οι αρχές στη χώρα απασχόλησης πρέπει να προσπαθήσουν να μάθουν τι γίνεται. Και πάντα ε, έρχονται μετά τα γεγονότα. Πρέπει να είναι εκ των προτέρων ενημερωμένοι στη χώρα απασχόλησης. Γι' αυτό θέλουμε υποχρεωτική εκ των προτέρων ενημέρωση ότι κάποιος πρόκειται να αποσπαστεί. Και αυτό που επίσης δεν υπάρχει είναι συγκεκριμένες και οδυνηρές σε κάποιες χώρες υπάρχουν. Αλλά τι γίνεται όταν οι εργαζόμενοι έχουν επανέλθει ήδη στη χώρα τους, πώς θα μπορέσουν να ζητήσουν να λάβουν αποζημιώσεις. Είναι πολύ περίπλοκη η κατάσταση. Στα χαρτιά μοιάζουν ωραίες αυτές οι διατάξεις, πώς ας πούμε να ξεκινήσουν ένδικες διαδικασίες, αλλά στην πράξη περισσότεροι εργαζόμενοι αποφασίζουν να μην ε, αρχίσουν ε, όλες αυτές τις ε, περίπλοκες διαδικασίες γιατί είναι ιδιαίτερα κανθόδης. Ποια είναι λοιπόν η πραγματικότητα. Υπάρχει σε μεγάλο βαθμό καταστρατήγηση της απόσπασης λόγω αυτοαπασχόλησης. Η όλη οδηγία μπορεί να καταστρατηγηθεί εάν κάποιος είναι ψευδός αυτοαπασχολούμενος. Πολύ αποσπασμένοι ξαφνικά υπογράφουν ένα κείμενο όπου αναφέρεται ότι ξαφνικά έχουν γίνει αυτοαπασχολούμενοι. Πολύ συχνά δεν ξέρουν ούτε καν τι υπογράφουν. Είναι γραμμένο το κείμενο σε γλώσσα που δεν καταλαβαίνουν. Και επειδή ε, του αρέσει ιδιαίτερα, είναι πολύ χαρούμενοι που βρήκαν ε, μια δουλειά στο εξωτερικό, υπογράφουν ό,τι να είναι. Επίση πολλά κείμενα αλλοιώνεται των υστέρων οι καταστάσεις ορών εργασίας, όλα αυτά αλλοιώνονται. Και αν υπάρχει επιθετητής εργασία, τους λένε ε, να κρυφτείτε, να σηκωθείτε τρέχοντας να φύγετε, να πείτε ψέματα ή θα τους δείξετε αυτό και το τάδε έγγραφο. Αυτές είναι οι πιο συνήθει συγκεκριμένε οδηγίες που λαμβάνουν. Συμπέρασμα. Η κατάχρηση των αποσπάσεων είναι η πραγματικότητα. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε. Πρέπει πολλά να κάνουμε. Χρειάζονται λύσεις στο επίπεδο των κρατών μελών. Σε ορισμένα κράτη-μέλη πρέπει να επιμείνουμε να υπάρχει σωστή εσωτερική προσπάθεια συντονισμού. Δεν υπάρχει ροή σε πολλές χώρες ε, πληροφοριών μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας, και τους ε, επιθεωρητές για θέματα μετανάστευσης. Οπότε δεν λειτουργεί αποτελεσματικά η διοίκηση της χώρας εσωτερικά. Είναι προφανές ότι οι υποχρεώσεις που υπάρχουν σε αυτή την οδηγία 91533 θα έπρεπε να εφαρμοστούν. Είναι απαράδεκτο η οδηγία αυτή που είναι ενισχύει εδώ και τόσα χρόνια να μην εφαρμόζεται στην πράξη αυτή η η οδηγία δεν εφαρμόζεται. Πρέπει να συζητήσουμε το γιατί δεν εφαρμόζεται. Ένα τρίτο πρόβλημα είναι η ενημέρωση. Είναι θέμα κλειδί. Η ενημέρωση πρέπει να είναι σαφής, απλή, προσβάσιμη. Πρέπει να τους χορηγείται πληροφόρηση για τις συνθήκες εργασίας που πρέπει να υπάρχουν, αυτό είναι ευθύνη των κρατών μελών, όπως σας είπα ήδη, στην πράξη αυτή η πληροφόρηση είναι ιδιαίτερα ανεπαρκής. Είμαι απόλυτα πισμένος ότι οι κοινωνικοί εταίροι, ιδιαίτερα στον τομέα των οικοδομών, θα ήταν διατεθειμένοι να χορηγήσουν αυτή την ενημέρωση, αλλά όλες οι προσπάθειες που έχουν επιτελεστεί μέχρι τώρα χρηματοδοτούνται από τους κοινωνικούς εταίρους. Αυτό είναι πολύ άκομψο, δεν είναι υποχρέωσή τους. Υπάρχει λοιπόν ε, καλή θέληση των κοινωνικών εταίρων να βοηθήσουν. Αλλά πρέπει και οι άλλοι να δώσουν κάτι. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η διαμεθοριακή συνεργασία. Ναι, ναι, θα, θα κλείσω εδώ. Θα κλείσω εδώ. μαζί με τους εργοδότες στον τομέα μας θεωρούμε ότι ένα καινοτόμο μέσο που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε είναι αυτή η πρώτερη υποχρεωτική ενημέρωση για τους εργαζόμενους που πρόκειται να αποσπαστούν ούτως ώστε στη χώρα απασχόλησης η επιθεώρηση εργασίας να γνωρίζει εκ των προτέρων πότε θα φτάσουν οι αποσπόμενοι αυτό θα διευκόλυνε τη δουλειά της επιθεώρησης εργασίας τρομερά. Πόσοι πρόκειται να αποσπαστούν, σε ποιο τόπο εργασίας, για πόσο χρονικό διάστημα. Κάτι άλλο που θα θέλαμε να προτείνουμε, πολύ καινοτόμο, αλλά όπως σας είπα υπάρχουν στις ε, γραπτές απαντήσεις μας. Υπάρχουν και άλλα λοιπόν, αλλά όπως σας είπα υπάρχουν γραπτές απαντήσεις μας και ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ και πυκνό. Ο επόμενος τώρα. Ε, ο καθηγητής Ιβ Ζόρενς στο Πανεπιστήμιο της, ε, του Γκέντ, ε, Ιστιτούτο Διεθνής Έρευνας στην τομέα της Απάτης, στην κοινωνικό τομέα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε κάποιες ιδέες σε σχέση με την πρόταση περιλοποίησης οδηγίας. Ε, η ομιλία μου θα διαρθρωθεί γύρω από τις ερωτήσεις ε, και θα μιλήσω πολύ για την ε, από κοινού και ισολόκληρον ευθύνη, διότι μόλις ολοκληρώσαμε μία μελέτη που μας ζήτησαν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για αυτό το ζήτημα. Το θέμα της υπεργολαβίας και της εξωτερικής ανάθεσης παίζουν ζωτικό ρόλο στην αγορά εργασίας πλέον σε τέτοιο βαθμό που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιστρέψουμε αυτή την τάση αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Δεν μπορούν να γίνουν δεκτές αυτές οι πρακτικές όταν οδηγούν σε παράκαμψη των νομικών διατάξεων. Ποιες είναι οι βασικές ατέλειες της νομοθεσίας για την προστασία των εργαζομένων. Είναι αυτές που σχετίζονται με την εφαρμογή ε, των διατάξεων σε σχέση με τις διαδικασίες επιθεώρησης διασυνοριακών ελέγχων και συνεργασίας των εποπτικών οργάνων Παρότι μιλάμε για ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων και υπηρεσιών, ε, είναι παράδοξο, αλλά δεν υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία των επιθεωρητών, ε, ούτε και ικανοποιητική ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτό καλύπτει όλα τα στάδια, από την επιθεώρηση μέχρι την επιβολή ε, ποινών. Ποιοι είναι βασικοί τρόποι παράκαμψη των ελαχίστων προτύπων χρησιμοποιείται το ότι δεν υπάρχουν ίσοι όρια ανταγωνισμού, υπάρχουν ψευδοαπασχολήσεις, η διασυνοριακή συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών είναι ατελής και ανύπαρκτες και αυτό είναι γενικώ γνωστό. Άρα είναι σχεδόν αδύνατο σε διασυνοριακό επίπεδο να εφαρμοστεί οποιαδήποτε απόφαση. Επίση, σε επίπεδο διοικητική και νομική ε, συνεργασία ε, επιδέχεται η διαδικασία βελτιώσει. Σήμερα ε, μπορούμε να βρούμε διάφορε αιτίε για αυτά τα φαινόμενα. Γλωσσικέ ελλείψει, έλλειψη γνώση για την κείμενη νομοθεσία του κράτου μέλου, το ότι αγνοούμε ποια είναι η αρμόδια αρχή, επιβολή διασυνοριακών προστήμων, εφαρμογή Τη απόφαση του Συμβουλίου σε σχέση με την αμοιβή αναγνώριση των χρηματικών πίνων που ισχύουν μόνο για τι διοικητικές που δεν ισχύει για τις διοικητικές κυρώσεις αλλά μόνο για τις ε, ποινικέ ε, κυρώσεις ε, καθυστερήσεις σε σχέση με την απόκτηση των απαιτούμενων πληροφοριών για τη διεξαγωγή ελέγχου κτλ. Λοιπόν, οι μηχανισμοί από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεωρούνται υπανάκια και μία από τις βασικές επικρίσεις που δέχεται αυτό το σύστημα είναι ότι ο ρόλος της επιθεώρησης έχει περάσει πλέον σε ιδιωτικές εταιρείες διότι και οι ίδιε οι αρχέ ε, ε, προσκρούν σε κολλήματα που δεν μπορούν να υπερπηδήσουν επίσης. Ε, ε, σε σχέση με την αποφυγή του αθέμητου ανταγωνισμού θεωρείται ότι ε, με το ισχύον ε, σύστημα της υπεργολαβίας γίνεται σωστότερη η επιλογή των υποψηφίων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το σύστημα έχει ισχυρή αποτρεπτική ισχύ για να αποφύγει κανείς την ευθύνη και προς συμφέρον του θα επιλέξει καλύτερους υπεργολάβους. Όμως στην πράξη δύσκολο μπορεί κανείς να επιβεβαιώσει αυτή τη θεωρία διότι όταν ε, ποσοστικοποιούμε τις πληροφορίες ε, για συγκεκριμένες ε, υποθέσεις που έχουν ρυθμιστεί για την αποκοινού και εις ολόκληρον ευθύνη είναι ελάχιστες και έχουμε ένα μάλλον περιορισμένο σύστημα απόδοσης ευθύνης και παρότι αυτά τα συστήματα εφευρέθηκαν για τη μαζική εισρωή αλλοδαπών εργαζομένων χρησιμοποιούνται σε χώριους και για εργολάβους που δραστηριοποιούνται ούτως ή άλλω ε, στο ε, εν λόγω κράτο μέλος. Οι ίδιοι εργαζόμενοι εξάλλου πρέπει να κινήσουν τη διαδικασία σε περίπτωση παραβίαση των δικαιωμάτων του ε, στην αλυσίδα υπεργολαβία. Και πολλοί εργαζόμενοι θεωρούν ότι δεν μπορούν να κινηθούν διότι φοβούνται τα αντίπεινα, παραδείγματο χάρη από τον εργοδότη ή από τι αρχέ, διότι δεν ενημερώνονται σωστά. Και εδώ θα μπορούσαμε να κρατήσουμε ένα σημαντικό ρόλο ενημέρωση. Σε πολλές ε, χώρες ε, φαίνεται ε, ότι τα συνδικάτα δυσκολεύονται να έρθουν καν σε επαφή με τους αλλοδαπούς εργαζομένους και όταν δεν απαιτείται δικαστική διαδικασία κινείται ταχύτερα η διαδικασία και μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι είναι θετική αυτή η εξέλιξη. Αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε σχετικά με το αν ένας μηχανισμός που λειτουργεί σε χώρο επίπεδο θα μπορούσε να μεταφερθεί αυτούς ή ως ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα στατιστικά δεδομένα στοιχεία που έχουμε από τη Γερμανία σε σχέση ε, με τις καταγγελίες ε, σε σχέση με τη χρονομίσθωση ε, παραθεριστικών κατοικιών μας δείχνουν ότι έχει χρησιμοποιηθεί το σύστημα για 200-300 υποθέσεις το χρόνο. Το ίμιση επιλήθηκαν εξοδικαστικά. Ε, και οι εισφορές σε αυτά τα ταμεία ανέρχονται σε 90 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2006 έως 2011. Τέτοιες εθνικές διατάξεις για την αποκοινού και ευθύνη δύσκολα είναι εφαρμοστές σε διασυνοριακές υποθέσεις και σίγουρα αυτό το επιχείρημα συνηγορεί υπέρ του ευρωπαϊκού συστήματος ε, ε, της αποκοινού και ευθύνη που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε διασυνοριακές υποθέσεις. Ασμένες χώρες έχουν ένα εναλλακτικό σύστημα, κυρίως στις σκανδιναβικέ ε, χώρες. Έχει δοθεί ένας πάρα πολύ σημαντικός ρόλος ε, στα συνδικάτα. Στη Σουηδία, Φερρυπίν, υπάρχει το δικαίωμα διαπραγμάτευση ε, και άρνηση κυρία των εργαζομένων για να μην εισέλθουν σε μια έκνομη σύμβαση απασχόληση. Όμως στην πράξη δεν χρησιμοποιούνται αυτέ οι διατάξει. Οι εργοδότες πάντως και τα συνδικάτα εισέρχονται σε διαπραγματεύσει. Στη Φινλανδία, δύο, ο πελάτης υποχρεούται να συλλέξει αποδείξει σε σχέση με την αξιοπιστία ενό υπεργολάβου προτού συνάψει τη σύμβαση και κοινωνικέ ρήτρε που υποχρεώνουν του υπεργολάβου να συμμορφωθούν με τι διατάξει περί συλλογικών αποζημιώσεων συμπεριλαμβάνονται μέσα στι συμβάσει. Επίση, υπάρχουν διάφορα εναλλακτικά μέτρα ενημέρωση που διευκολύνουν την παρατήρηση και την εποπτεία όπω παραδείγματο χάρη ε, τα, ε, ε, μηχανισμοί πρώτερης κοινοποίησης ε, που χρησιμοποιούνται σε 18 κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θεωρείται ότι η κοινοποίηση είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την ενημέρωση και τη, σχετικά με τη δραστηριοποίηση αλλοδαπών εταιριών ε, στην επικράτεια ενός κράτου μέλους. Πάντω, το βελγικό σύστημα βρίσκεται πρώτων δικαστηρίων και αν πιστέψουμε τον Γενικό Εισαγγελέα, πόρο απέχουμε από την επίλυση τη υπόθεση Για την ευθύνη τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν αυτό το σύστημα θα περιοριστεί σε διασυνοριακέ υποθέσεις, δεν υπάρχει κανένα τεκμήριο ότι αν εισαχθεί αυτό το σύστημα μόνο για διασυνοριακές υποθέσεις, αυτό δεν θα μας οδηγήσει σε περιορισμό της αγοράς εργασίας του κράτου μέλους υποδοχής. Ε, οι και κυρίω μικρομεσαίες θα το σκεφτούν δις ε, πρωτού κάνουν κάτι τέτοιο και πιστεύω ότι ένας παίκτης της αγοράς ε, μπορεί ε, πολύ εύκολα να ε, παρακάμψει ε, ε, τις διατάξεις ενός τέτοιου συστήματος για την απόδοση ευθύνης, διότι γνωρίζει καλύτερα την εγχώρια κατάσταση. Τώρα, αν θα διευρυνθεί το σύστημα στους παρόχους υπηρεσιών, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτό περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών. Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι θα πρέπει να αιτιολογούμε την αίτηση περί κοινοποίησης. Σας παραπέμπω στην ομολογία του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχολιάζει την αιτιολόγηση και την θεωρεί επιπρόσθετη υποχρέωση. Ο Ευρωπαίος νομοθέτης θα πρέπει να έχει μεγαλύτερο περιθώριο ερμηνείας ε, για το θέμα της αιτιολόγησης. Ε, όμως ε, δεν αποκλείω να ανακάμψει αυτό το θέμα ενώπιον του Δικαστηρίου της Ένωσης, διότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν παρεμφερείς κανόνες για να ρυθμίσουν όμως αμυγός εθνικές καταστάσεις. Και όταν λειτουργούν οι εταιρείε καλή την πίστη. Ε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ε, όμως υπάρχει μία αμφισημία, ε, διότι η προληπτική εποπτεία σε συνδυασμό με την από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη δημιουργούν προβλήματα παρότι υπάρχουν λόγοι που αιτιολογούν μια τέτοια κίνηση. Έχουμε την οδηγία 2952 για τους παράνομα απασχολούμενους και εκεί υπάρχει σχετική διάταξη για την προληπτική εποπτεία και και ε, αναφέρεται ότι όσοι ε, ε, συμμορφώνονται με αυτήν την διάταξη απεκδίονται αυτήν την από κοινού και ισολόκληρον ευθύνη και είναι πάρα πολύ εύκολο κανείς να αντιγράψει το κείμενο της οδηγίας και να παρακάμψει έτσι το σύστημα. Συνοψίζοντας θα ήθελα να πω ότι οποιοδήποτε σύστημα ευθύνης δεν μπορεί να αντικαταστήσει ε, την έλλειψη δράσης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη γενικότερη ρύθμιση της αγοράς. Έλλειψη ε, ε, επιπρόσθετων μέτρων δεν θα επαρκέσει η εισαγωγή αυτού του συστήματος για την πρώτερη κοινοποίηση, παραδείγματος χαρήν. ενημέρωση σε διασυνοριακές υποθέσεις, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διοικητικών αρχών, βελτίωση της διασυνοριακής εφαρμογής αποφάσεων ποινικού και διοικητικού χαρακτήρα, επιβολή ε, ποινών, ζητήματα όπως ε, η παραβίαση των δικαιωμάτων των νομικών ε, προσώπων και τέλος, αλλά και σημαντικό το θέμα των ψευδοαπασχολούμενων δεν λύνονται μόνο με αυτό το σύστημα της αποκοινωνικής ολόκληρων ευθύνη. Αυτό το φαινόμενο των ψευδοαπασχολούμενων μόνο θα εξαπλωθεί αν δεν λάβουμε πρόσθετα μέτρα. Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε τη σημασία αυτού του φαινομένου. Σας ευχαριστούμε. Ήταν από διαφορετική από την γωνία. Ο κύριος Στίγ Νόργαρντ είναι ανώτερος σύμβουλος στο Υπουργείο Εργασίας της Δανίας. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ. Είναι μεγάλη τιμή να είμαι ενώπιόν σας, στην Επιτροπή σας Δέκα λεπτά είπατε. Μερικά θέματα για το δανέζικο σύστημα και μερικά γενικότερα. Αρχίζω με το ερώτημα που θεωρώ ότι είναι ο κυριότερος τρόπος για την παράκαμψη των ελαχίστων προδιαγραφών, γιατί είναι βασική αυτή η αντιμετώπιση. Στη Δανία δεν έχουμε υποχρεωτικά μίνιμουμ για την αμοιβή, δεν έχουμε ούτε νομοθεσία, ούτε ε, σφαιρικά, σφαιρικές συλλογικές συμβάσεις. Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να καταλήξουν στις συλλογικές συμβάσεις στη τελευταία ανάλυση και μέσω συλλογικής δράσης ενδεχομένω Η Δανία και η Σουηδία έχουν κάποιες ομοιότητες. Οι αρχές ε, είναι ίδιες στις δύο χώρες. Όταν μιλάμε για αμοιβή, το πρόβλημα δεν είναι το θέμα μη εφαρμογή ενό ελάχιστου μισθού, αλλά πώς να καθορίσεις ε, τις μίνιμουμ αποδοχές, γιατί μιλάμε για ξένες εταιρείε. Οπότε τα συνδικάτα έχουν πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσουν λόγω της προσωρινής ε, και σύντομης παρουσίας των αποσπασμένων. Δύσκολα λοιπόν ε, βρίσκεις αυτές τις εταιρείε και έρχεσαι σε επαφή μαζί τους. Αλλά και αν υπάρξει συμφωνία, υπάρχουν πολλά προβλήματα καταστρατήγησης, γιατί τα συνδικάτα έχουν δει πόσο δύσκολο είναι, έχουν διαπιστώσει, πόσο δύσκολο είναι να λάβουν συντροματικές πληρωμές που δεν έχουν δοθεί από τις χώρες προέλευσης, παρά το ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά μέσα. Πώς λοιπόν καταφέρνει κανείς να βρει ποιες είναι αυτές οι ξένες εταιρείες να έρθει σε επαφή μαζί τους. Το 2008 Έχουμε ένα σύστημα ενημέρωσης για τους ξένους εργαζόμενους. Έτσι είναι πιο εύκολο για τα συνδικάτα να επικοινωνήσουν με τις ξένες εταιρείε. Αλλά επίσης βοηθάει και την ε, επιθεώρηση ε, για λόγους υγείας και ασφάλειας τοποεργασίας για να μπορούν να κάνουν ελέγχους. Με βάση την ανακοίνωση του 2006 της Επιτροπής εισαγάγαμε αυτό το σύστημα και με βάση την ομολογία του δικαστηρίου. Και έχει γίνει πρόταση να συμπεριληφθεί στο άρθρο 9 αυτής τη οδηγίας επιβολή τώρα, τη νέα οδηγία. Υπάρχει υπηρεσιών, πρέπει να δώσουν το όνομα της εταιρεία, τη διεύθυνση, άλλες πληροφορίες ε, πού ακριβώς θα δοθούν ε, οι υπηρεσίες, ε, πόσο θα κρατήσει η απόσπαση, το όνομα των αποσπασμένων και ένα άτομο επαφή. Αυτές οι πληροφορίε πρέπει να μπουν ηλεκτρονικά απευθεία Αυτό σημαίνει ότι είναι εύκολο να στείλεις και στις υπηρεσίες τα στοιχεία αυτά που ελέγχουν αν έχει υπάρξει αυτή η πρώτερη ενημέρωση. Αυτή η υποχρέωση είναι καινούρια, δεν ήταν εξ αρχής ε, υποχρεωτική. Διαπιστώσαμε όμως ότι πολλές φορές υπάρχουν υπηρεσιών δεν έστελναν την ενημέρωση των προτέρων. Έτσι λοιπόν οι Δανείοι ε, διασφαλίζουν κοινή ευθύνη με ρωτήσανε εάν αυτό το σύστημα πρώτερης ενημέρωσης μπορεί να έχει να κάνει με το σύστημα κοινών υποχρεώσεων. Όπως είπα και κάποια κράτη-μέλη έχουν τέτοια συστήματα. Ε, ακόμη και χώρες που έχουν κοινή, ε, υποχρεώσεις. Η λογική αυτών των χωρών είναι ότι το σύστημα κοινή υποχρέωση είναι μόνο ένα δίκτυο ασφαλείας. Σε πρώτη φάση, στόχος μας είναι ο πάροχος υπηρεσιών να πληρεί τις υποχρεώσεις του και να ενημερώνει για τους ε, προς απόσπαση. Φυσικά, ένα τέτοιο σύστημα κοινή ε, υποχρέωση θα μπορούσε να συνδυαστεί με το δικό μας σύστημα. Θα είχε έννοια λοιπόν οι υποχρεώσει των παρόχων να βάλουν τα στοιχεία στο σύστημά μας που λέγεται root θα μπορούσε να θεωρηθεί και επαρκή επιμέλεια με την έννοια της πρότασης της οδηγίας όπως είναι τώρα. Κάτι προσωπικό τώρα. Όταν υπάρχει σύστημα κοινών υποχρεώσεων, υποχρεώνει αυτόν που λαμβάνει τι υπηρεσίε να κάνει και αυτό κάποιου ελέγχου. Αυτό είναι ο στόχο. Αυτό που λαμβάνει λοιπόν υπηρεσίε μπορεί να πάρει προφόρηση που οι αρχέ τη χώρα υποδοχή δεν μπορούν εκ των προτέρων να ζητήσουν για την καλή συμπεριφορά, για παράδειγμα, του παρόχου. Αλλά οι λήπτε των υπηρεσιών θέλουν αυτέ τι προφορίε για να μην ε, έχουν ευθύνη μετά. Αν υπάρχει λοιπόν ένα κεντρικό μητρό όπου θα μπορούσαν να εγγραφούν εταιρείε μόνο εφόσον πληρούν τις υποχρεώσεις του στο κράτος προέλευσης, δεν, χρειαζόμαστε, δεν θα χρειαζόμαστε αυτό το σύστημα ε, ε, κοινών υποχρεώσεων και επαρκούς επιμέλειας. Ο λήπτης θα έβλεπε εάν ο πάροχος είναι στο Μητρό. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι οι αρχές του κράτους ε, προέλευσης θα είχαν περισσότερε υποχρεώσει, αλλά θα διασφάλιζε για πραγματικέ εταιρείε πραγματική κινητικότητα των εργαζομένων. Και ούτε θα χρειαζόταν οι αρχέ να απευθύνονται μία στην άλλη από χώρα σε χώρα, αλλά βεβαίω είναι ίσω ιδιαίτερα φιλόδοξο αυτό που προτείνω. Σω δεν μπορεί να γίνει στα πλαίσια αυτή τη οδηγία επιβολή. Είναι μακροπρόθεσμο στόχο. Τέθηκε επίση το ερώτημα, ένα κεντρικό σύστημα εγγραφή πώ θα γίνει. Χρειαζόμαστε ένα κεντρικό οργανισμό γι' αυτό, ευρωπαϊκό ή μέσω διμερού συνεργασίας. Έχουμε το σύστημα για ανταλλαγή πληροφοριών που χειρίζεται η μεσω διμερου συνεργασια Επιτροπή για κοινωνικούς, κοινωνικές πληροφορίες. Θα μπορούσαμε να έχουμε και διμερή συνεργασία, αλλά οι χώρε που διμερώ συνεργάζονται θα πρέπει να ορίσουν κάποια αρχή σε μία από τι δύο χώρε για να είναι υπεύθυνη για αυτήν την ανταλλαγή πληροφοριών. Γι' αυτό το μητρό, α πούμε. Υπόθηκε ότι το σύστημά μας είναι ευρύτερο σε πεδίο εφαρμογή από ένα απλό μητρό. Αυτό ίσως έχει να κάνει με το ότι οι ξένες εταιρείε πρέπει να, προφορήσουν και, να δώσουν προφορίες και για τον τόπο εργασία κτλ. Αλλά αυτό είναι με βάση και τους προσανατολισμούς του άρθρου 9. Και, έχει γίνεται και αυτό γίνεται και σε άλλου τομεί, για παράδειγμα, παροχή υπηρεσιών. Πρέπει να μπορούν να αποδείξουν, για παράδειγμα, ότι πληρώνουν τι κοινωνικέ ασφαλίσει. Άρα πρέπει να ενημερώσουν για τον τόπο εργασία. Λογικό να ενημερώσουν για τι εγκαταστάσει του τόπου εργασία, γιατί οι αρχέ πρέπει να κάνουν ελέγχου. Πρέπει να ξέρουν πού είναι ο τόπο εργασία. Στι παρατηρήσει επίση λέγεται ότι αυτά που έχουμε στο σύστημά μα το root, είναι ανακριβή. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι πολύ δύσκολο να ε, εφαρμόσουμε παντού τις ίδιες αρχές και τις ίδιες διαδικασίες. Όταν το root το εισαγάγαμε, το ελέγξαμε και με ξένους χρήστες. Τους ρωτήσαμε αν είναι σαφή τα πράγματα, αλλά παρόλα αυτά, παρόλους αυτούς τους ε, εισαγωγικούς ελέγχους, υπάρχουν ε, ανακρίβες και χρειαζόμαστε πολλές φορές επαφές με άλλες χώρες για να διευκρινιστούν θέματα. Πώς θα είμαστε λοιπόν σίγουροι ότι όλη η πληροφόρηση είναι μεταφρασμένη. Η απάντηση είναι ναι με το προβλέπει το άρθρο 5 αλλά δεν ξέρω αν αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Γιατί ελπίζω όλη η πληροφόρηση να είναι σχετική και η ίσως να μην είναι μάλλον ε, σχετική όλη η πληροφόρηση, οπότε να μεταφράζονται όλα όσα είναι στο μητρό μας, στο σύστημά μας, σε όλες τις γλώσσες θα ήταν ίσως υπερβολικό. Πρέπει να είναι πιο στοχευμένη η χορήγηση πληροφοριών στις ξένες εταιρείε. Το θέμα αυτό βεβαίως μας ενδιαφέρει και για την οδηγία για τις υπηρεσίες. Η ανακοίνωση της Επιτροπής τον Ιούνιο καταδεικνύει ότι δεν λειτουργεί πάντα το ενιαίο σημείο επαφής όπως θα ελπίζαμε. Τώρα μια ερώτηση για το άρθρο 9. Εάν δηλαδή λόγω τη διαφορετικότητα των μηχανισμών ελέγχου, πώ θα συνεχίσουν του εθνικού ελέγχου του αποτελεσματικά τα κράτη-μέλη με βάση τη νέα οδηγία επιβολή. Πιστεύω ότι η πρόθεση τη επιτροπή είναι να εδρεώσει, μάλλον να βασιστεί στην ομολογία για να εδρεώσει το νέο σύστημά τη. Αλλά μ, υπάρχουν αμφισβητήσει γι' αυτό. Κάποια κράτη-μέλη, όπω η δική μου, όπω το δικό μου κράτο μέλο, πιστεύουν ότι χρειάζεται ευελιξία για το μέλλον για περιπτώσεις που δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Αν βασιστούμε μόνο στο άρθρο 9, μπορεί να έχουμε κατόπιν ε, προβλήματα στην εφαρμογή και δικαστικές ε, αμφισβητήσεις. Υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές από κράτη-μέλη που περιορίζονται λόγω της νομολογίας του δικαστηρίου ή απαγορεύονται πλέον. Αναφέρθηκε το θέμα των ψευδώς ε, αυτοαπασχολουμένων που καταστροτηγεί την οδηγία. Το Βέλγιο προσπάθησε να εισαγάγει και τους αυτοαπασχολούμενους στο σύστημα Μιμόζα, αλλά η Κομισιόν ε, το αμφισβητεί στο δικαστήριο. Ας περιμένουμε λοιπόν την απόφαση του δικαστήριου σε δύο-τρει μήνες. Χρειάζεται επίσης, ε, ρωτήθηκα, ευρωπαϊκό νομοθέτημα για την εφαρμογή των ελάχιστων προδιαγραφών όπως προβλέπει η οδηγία. Νομίζω ότι μακροπρόθεσμα θα μπορούσαμε να επιτύχουμε τους στόχους ε, για τους οποίους πρώτο βήμα είναι αυτή οι πρώτες οδηγίες, ώστε να μην υπάρχουν ψεύτικες εταιρείες, ψεύτοεταιρείες. Πολλά προβλήματα προκύπτουν επειδή κάποιες εταιρείες έχουν εταιρείε βίο ή είναι και εντελώ ε, Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ και σας. Ε, φτάσαμε τώρα στον τέταρτο εμπειρογνώμονά μας, τον κύριο Τόμας Λάιχερ, που είναι Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Οικοδομικών Επιχειρήσεων. Ε, και η ομιλία του έχει ήδη διανεμηθεί στα μέλη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Απασχόλησης για τη διοργάνωση της σημερινή ακρόασης και επίσης η ΦΙΕΚ έχει την ευκαιρία να ε, εκθέσει την κατάσταση ως προς τις οικοδομικές επιχειρήσεις. Είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Οικοδομικών Εταιριών, η ΦΙΕΚ, και εκπροσωπεί 33 εθνικές ενώσεις από 29 διαφορετικές χώρες. Εκπροσωπούμε οικοδομικές επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, από τη μικρή, μεγάλη πολυεθνική συμπραξία μέχρι και τη μικρή οικογενική ε, επιχείρηση. Όλες δραστηριοποιούνται εδώ στον κατασκευαστικό τομέα. Ε, επίσης εκπροσωπούμε τους εργοδότες ε, στον κλαδικό ευρωπαϊκό διάλογο για τον κατασκευαστικό τομέα. Θα ήθελα τώρα να επικεντρώσω την προσοχή μου στα συγκεκριμένα ερωτήματα που μας υποβάλλατε. Θα ήθελα βεβαίως ε, να σχολιάσω και κάποια άλλα ζητήματα και να αναπτύξω περαιτέρω τα ερωτήματά σας αργότερα, αν το επιθυμείτε. Πρώτον, ποια μέτρα θα πρέπει να αναλάβουν τα κράτη-μέλη, ούτω ώστε ε, να υπάρξει συμμόρφωση με τι διατάξει αυτή τη οδηγία. Ένα από τα στοιχεία κλειδί για την ορθή εφαρμογή τη οδηγία περί απόσπαση είναι η διαθεσιμότητα των πληροφοριών οι πληροφορίες, ενημέρωση μάλλον των επιχειρήσεων, ώστε να γνωρίζουν ποιες διατάξεις καλούνται να εφαρμόσουν και ενημέρωση των εργαζομένων για να γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματά τους. Ενημέρωση επίσης των δημοσίων αρχών, ούτως ώστε να μπορέσουν να ελέγξουν την εφαρμογή ε, της σχετικής νομοθεσίας. Η οδηγία περί απόσπασης ενέχει κάποιες ε, θετικές διατάξεις, ε, αλλά χωλαίνει και σε κάποια σημεία και επιδέχεται βελτιώσεις. χάρη, ε, για να ε, καταστούν δυνατή αποτελεσματική έλεγχοι, οι αρμόδιε εθνικές αρχές ε, θα πρέπει εγκαίρω να ενημερώνονται προτού αρχίσει η απόσπαση του εργαζομένου προτού ή προτού έρθει ένας αλλοδαπός πάροχος υπηρεσιών στην επικράτεια του κράτους. Ε, υπάρχουν φόβοι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη το κοινό αίτημα των κοινωνικών εταίρων από το κατασκευαστικό τομέα ε, FIAC WW. Ε, πιο συγκεκριμένα ζητήσαμε όλα τα κράτη-μέλη να έχουν ένα υποχρεωτικό σύστημα ενημέρωσης σε προτού η ίδια η απόσπαση με ποιο τρόπο μπορούμε να οργανώσουμε αποτελεσματικού ελέγχους όταν ε, οι δημόσιε αρχές δεν έχουν τόσο βασικές πληροφορίε. Από την εμπειρία μας ε, ε, που εφαρμόζονται, σε ποιο τομέα παρατηρούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα. Ε, συστηματικά ε, ε, προκύπτουν προβλήματα σε σχέση με την εφαρμογή σε κάποιες περιπτώσεις. Θεωρούμε ότι είναι δυνατή η ορθή εφαρμογή της οδηγίας πρώτον όταν είναι ξεκάθαρη η εφαρμοστέα νομοθεσία και είναι όλοι απολύτως ενημερωμένοι. Δεύτερον, υπάρχει λεπτομερής ενημέρωση και για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζομένους σε σχέση με την εφαρμοστή νομοθεσία για να κατανοήσουν ότι είναι προς συμφέρον τους. Επίσης, πέρα από την διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων, οι επιθεωρητές θα πρέπει να έχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες και τα απαιτούμενα μέσα για να διεξαγάγουν ε, τον έλεγχο. Φοβούμαστε και πιστεύουμε ότι η προτινόμενη οδηγία δεν καλύπτει πλήρω ε, όλα αυτά τα προαναφερθέντα κριτήρια. Ποια είναι τα μέτρα λοιπόν που πρέπει να αναλυθούν. Στα περισσότερα κράτη-μέλη υπάρχουν διάφορε πηγέ ενημέρωση σε σχέση με την απόσπαση γενικότερα, αλλά η επιχείρηση χρειάζεται και πρακτικέ πληροφορίε, εύληπτε πληροφορίε ε, που ε, σχετίζονται με την δραστηριότητά τη. Η διαθεσιμότητα τέτοιων πληροφοριών σε διάφορε γλώσσε είναι επίση μια σημαντική διάσταση του ζητήματο. Γι' αυτό το λόγο μεταξύ άλλων το 2009 αναπτύξαμε και δρομολογήσαμε μαζί με του συναδέλφου μα από τα συνδικάτα μια κοινή ιστοσελίδα σε σχέση με την απόσπαση στον κατασκευαστικό τομέα. Αυτή η ιστοσελίδα προέκυψε από, από δύο ανεξάρτητε μελέτε, ότι είναι παράδειγμα βέλτιστη πρακτική. Ω προ την προσβασιμότητα, ή μάλλον ως προς την αδυναμία πρόσβασης ε, στις απαιτούμενες πληροφορίες. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Εγώ μελέτησα τις διατάξεις ε, της νομοθεσίας ε, με τις οποίες καλούμε, είμαι μάλλον να συμμορφωθώ είτε πρόκειται για την χώρα όπου διαμένω ή τη χώρα όπου θα εργαστώ προσωρινά. Οι αρμόδιες διοικητικές αρχές φέρουν το φορτίο, την υποχρέωση γνώμη της ενημέρωσης οι ευθύνες είναι ξεκάθαρες. Η, ακόμη και αν ε, κάποια στιγμή αλλάξουν αυτές οι διατάξεις, ε, μπορώ να προσαρμοστώ, εάν όμως είμαι ενημερωμένος για την αλλαγή. Όμως, αν ενημερωθώ μεταγενέστερα, μετά δηλαδή την αλλαγή, η αρχή που υποχρεούται να μου προσκομίσει τις πληροφορίες είναι εκείνη που πρέπει να υποστεί τις επιπτώσεις. Ε, τώρα οι υπηρεσίες προσωρινής απασχόλησης ε, πώς σχετίζονται με αυτό το φαινόμενο της απόσπασης. Τα ε, τα γραφεία εξέβρεση προσωρινής εργασίας δραστηριοποιούνται στα περισσότερα κράτη-μέλη και υπάρχουν δύο ευρωπαϊκά νομοθετήματα που καλύπτουν την προσωρινή απασχόληση. Η οδηγία περί απόσπασης και η οδηγία για τα γραφεία εξέβρεση προσωρινής απασχόλησης. Είναι αλληλοσυμπληρούμενε αυτέ οι οδηγίε και αλληλοενισχύονται ε, ως προς τις εφαρμοστέ διατάξεις, κυρίως ε, δε ε, για τις συνθήκε εργασίας. Τα περισσότερα κράτη-μέλη εφαρμόζεται η νομοθεσία της χώρα υποδοχή για τους εργαζομένους που έχουν σύμβαση απασχόληση με ένα γραφείο εξέβρεση προσωρινής εργασία. Ποιες είναι οι διατάξεις μας ρωτάτε που χρειάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ούτως ώστε να αποφύγουμε την ε, ε, υπόθεση Λαβάλ στη Σουηδία. Για την ε, υπόθεση Λαβάλ νομίζω ότι έχουμε πει τα πάντα ήδη, διείστανται οι απόψεις εξαρτάται αν εξετάζει κανείς το θέμα από την οπτική γωνία των ε, ε, εργοδοτών ή των συνδικάτων. Και οι πλέον επιφανείς νομομαθείς ε, έχουν διαφορετικές απόψεις. Εγώ δεν θέλω να ξεκινήσω νέα συζήτηση για αυτό το θέμα. Η ΦΙΑΚ πιστεύει ότι ακόμη και μετά την υπόθεση Λαβάλ και οι υπόλοιπε υποθέσεις που έχουν δικαστεί στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου θεωρούμε ότι αυτή η οδηγία είναι το κατάλληλο εργαλείο τόσο να κατοχυρωθεί η ελευθερία παροχής υπηρεσιών και η προστασία των δικαιωμάτων δικαιωμάτων των εργαζομένων. Δεν ε, χρειάζεται να τροποποιηθεί η πρόταση οδηγία. Καλωσορίζουμε δε το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προτείνει τώρα ε, η νέα τη πρόταση να συμπεριληφθεί σε ένα νέο σχέδιο περί εφαρμογή και σωστή μεταγραφή τη οδηγία για την απόσπαση. Σε σχέση τώρα με την παράκαμψη τη οδηγία. ο ευκολότερο τρόπο είναι αυτό το φαινόμενο τη της αυτοαπασχόληση. Το 2009 με του συναδέλφου μας από τα συνδικάτα ολοκληρώσαμε μία μελέτη για αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα και εκδώσαμε κοινέ ακατευθυντηρίες σε γραμμές. Είναι περίπλοκο το ζήτημα και ε, το εργασιακό δίκαιο, οι φορολογικέ ε, διατάξεις και άλλα τέτοια περίπλοκα εθνικά ζητήματα εμπλέκονται στην υπόθεση και σίγουρα υπερβαίνουν την απλή απόσπαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, γι' αυτό το λόγο δεν ε, προσπαθεί να ρυθμίσει το πρόβλημα μέσα στην ε, πρόταση αυτή νομοθετικού περιεχομένου. Όμως κάποια από τα προβλήματα που συνδέονται με την απόσπαση σίγουρα μπορούμε να τα εξετάσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιληφθεί αυτών των ζητημάτων. Εφιστάμενε βέλτιστε πρακτικέ. Η επόμενη ερώτηση. Κατάλληλοι έλεγχοι και μηχανισμοί παρακολούθηση, αποτελεσματικέ επιθεωρήσει και έλεγχοι απαιτούνται ούτω ώστε να είναι ίση η ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις και να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των εργαζομένων. Όμω οι διατάξει που μα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μα προτείνουν έναν ολοκληρωμένο κατάλογο διοικητικών υποχρεώσεων και μέτρων ελέγχου που θα μειώσουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα διεξαγωγή ελέγχων. Σε σχέση με την σημερινή κατάσταση, ένα τέτοιο περιορισμό δεν θα επιτρέψει την ορθή εφαρμογή, μεταφορά και εφαρμογή τη οδηγία απόσπαση και αντιβαίνει στον βασικό δεδηλωμένο στόχο τη οδηγία. Οι διατάξει αυτές υπερβαίνουν την ομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε σημαντικό βαθμό ε, θα ε, περιστήλουν τη δυνατότητα ελέγχου των αρμοδίων ε, αρχών γνωρίζουμε ότι ε, συμφωνούμε επ' αυτού με τους ε, συναδέλφους που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους. Ε, αν αυτή η πρόταση για την εφαρμογή της οδηγίας τροποποιηθεί καταλήλως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τρόπο ώστε οι απαιτούμενε πληροφορίες να είναι διαθέσιμες για τις επιχειρήσεις, για τους εργαζομένους και για όλους όσους καλούνται να διεξαγάγουν τους ελέγχους, αν έχουμε ένα αποτελεσματικό ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στις αρμόδιες εθνικές διοικητικές αρχές, σε αυτή περιπτώσει περιπτώσει όντω μπορούμε να επιτελέσουμε αποτελεσματικού ελέγχου ε, και να επιτύχουμε μια ε, διασυνοριακή εφαρμογή των αποφάσεων ε, περί χρηματικών και άλλων ποινών και προστήμων. Στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση με την τωρινή κατάσταση. Τα συμπεράσματά μου. Απήντησα στι ερωτήσει που με υποβάλλατε. Πρωτού όμω ολοκληρώσω την παρέμβασή μου, θα ήθελα να πω κάποια λόγια για το πλέον ακαθόδε ζήτημα του τεστ το θέμα της ε, κοινή ευθύνης. Η ΦΙΑΚ ε, δεν είναι κατά των συστημάτων κοινή ευθύνης, αυτά καθ' αυτά. Ε, υφιστάμενα τέτοια συστήματα που έχουν εφαρμοστεί στον κατασκευαστικό τομέα είναι από αντικείμενο διαπραγματεύσει ανάμεσα στου κοινωνικού εταίρου. Είμαστε κατά όμω τη ευρωπαϊκή παρέμβαση για το θέμα τη κοινή ευθύνη. Οι προτινόμενε διατάξει, κατά τη γνώμη μα, υπερβαίνουν την απλή εφαρμογή τη οδηγία για την απόσπαση, διότι στην πράξη οδηγούν σε ρύθμιση τη υπεργολαβία η εφαρμογή στις δραστηριότητες απόσπασης ε, συνιστά μεσοκόλλημα για τους αλλοδαπούς παρόχους υπηρεσιών διότι de facto ε, θα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αυτοί που θα θέλουν να χρησιμοποιήσουν αλλοδαπούς παρόχους υπηρεσιών εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο σύστημα ε, στο κράτος μέλος, συγκεκριμένα σε 16 από τις 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα από τα υφιστάμενα συστήματα κοινή ευθύνη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ξαναλέω εδώ ότι είναι προϊόντα των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στου κοινωνικού εταίρου και συνιστούν λεπτότατες ισορροπίε και ενδέχεται να ανατρέψουν τις σχέσεις ανάμεσα σε όλους του παραγωγικούς φορείς. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το θέμα ε, είναι και πρέπει να παραμείνει ε, ε, εθνικής Σα Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ για την συμβολή σα. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή εικόνα ως βάση για τη συζήτησή μας και για ερωτήσεις. Καλό λοιπόν τώρα τα μέλη της Επιτροπής μας να κάνουν ερωτήσεις. Έχουμε περιορισμένο χρόνο, οπότε θα ήθελα παρακαλώ δύο λεπτά να ομιλητή. Οι συνάδελφοι Κρίστενσεν και μετά Σλούτερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές μας ε, για τις ε, παρουσιάσεις που μας έκαναν. Εάν δούμε πώς έχει κατάσταση σε αρκετά μέλη κυρίως ας πούμε με τους μεταφορείς, ε, με πάρα πολλούς εργαζόμενους που είναι αποσπασμένοι αλλά που δεν καλύπτονται από την οδηγία αυτή για την απόσπαση των εργαζομένων. Ε, τι έγινε, πώς μπορεί κανείς να δώσει τη μάχη του κατά του κοινωνικού αυτού dumping και ειδικότερα στον τομέα των μεταφορών. Το άρθρο 3 μήπως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν μηχανισμός ελέγχου, δεν ξέρω αλλά μήπως θα μπορούσαμε να ζητήσουμε ένα έντυπο για μια υποχρεωτική δήλωση για την απόσπαση ορισμένων εργαζομένων. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, θα πρέπει να είμαστε υπέρ της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Τώρα το άρθρο 12, το άρθρο 12 για την ε, κοινή ευθύνη στη νέα οδηγία. Εκεί καλύπτονται μόνο λίγοι τομεί ε, όπως των οικοδομών. Πώς μπορούμε να έχουμε μια επέκταση και σε άλλους τομείς. Ε, και να μην ξεχνάμε ότι η ελεύθερη κυκλοφορία σε μερικές περιπτώσεις δεν επιτρέπεται ουσιαστικά και όταν υπάρχει μια απόσπαση βλέπουμε ότι παρακάμπτουν τα ισχύοντα. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Διάφορες ερωτήσεις έχω. Η πρώτη αφορά τον κύριο Μπίλεν από την Ομοσπονδία των Εργαζομένων στις Οικοδομές και το Ξύλο Έχω μπροστά την γραπτή σας απάντηση. Κάνετε σαφή έκκληση για να υπάρχει στην οδηγία επιβολής ορισμός του τι σημαίνει απόσπαση. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί θέλετε να υπάρχει τέτοιος ορισμός. Δεύτερη ερώτηση. Προς τον εκπρόσωπο από τη Δανία η εντύπωσή μου ε, είναι ότι είστε ευχαριστημένοι με το άρθρο 9. Με εκπλήσει αυτό. Διότι πρέπει να δούμε επίσης ότι το άρθρο 9 που μπαίνει τώρα αντί του άρθρου 5 της αρχικής πρότασης είναι πολύ πιο περιοριστικό και μειώνει τις δυνατότητες αποφασιστικών ελέγχων από πλευρά των κρατών μελών στα εθνικά του συστήματα. Αν διαβάσουμε επακριβώς το άρθρο 9. Γιατί ε, σας αρέσει τόσο πολύ το άρθρο 9 αν σας κατάλαβα καλά, είπατε ότι είναι καλό. Παρακαλώ, εξηγήστε μας. Γιατί και ποια είναι η πείρα από το πολύ επιτυχημένο δικό σας σύστημα. Προς ε, τον κύριο Σλάχερ, θέτω το ερώτημα. Είπατε ότι εάν υπάρχει καλή συνεργασία κοινωνικών εταίρων, μπορούμε να δημιουργούμε συστήματα που να είναι σχετικά αποτελεσματική έλεγχη και που επίσης, διασφαλίζουν δίκαιο ανταγωνισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα των υπηρεσιών. Μπορείτε να μας εξηγήσετε άλλη μια φορά κατά τη γνώμη, μας, κατά τη γνώμη σας, ανεξάρτητα από το κείμενο της Επιτροπής, τι συστήματα χρειαζόμαστε για να υπάρχει αποφασιστικός, αποτελεσματικός έλεγχος. Είπατε χρειάζεται ενημέρωση, ανταλλαγή προφοριών, αλλά υπάρχουν και σε κάποια κράτη μέλη συστήματα που να είναι λειτουργικά. Και πώς βλέπετε τους περιορισμούς που ε, εισάγει το άρθρο 9 της Κομισιόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και τους προσκεκλημένους μας. Κάτι που δεν καταλαβαίνω είναι πώς έχουν ακριβώς οι ορισμοί. Με δυσχεραίνει. Είναι πρόκληση. Γιατί εάν είναι περιοριστικοί οι ορισμοί, μπορεί να προκύψει μια κατάσταση όπου εξαιρούνται κάποιοι εργαζόμενοι και να αυξήσετε την ε, καταστρατήγηση. αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την απασχόληση, τις αποσπάσεις, την αυτοαπασχόληση, τις αποσπάσεις, Πώς θα διασφαλίσουμε την προστασία των εργαζομένων. Ίσως να φασιστούμε απλώς στην ίση μεταχείριση ως ε, λύση ανάγκης. γιατί έχουμε διαφορετικούς ορισμούς. Έχουμε την απόσπαση, έχουμε προσωρινούς εργαζομένους και τους κανονικούς εργαζομένους. Και παρεμβαίνει και η Ρώμη 1. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα των ψεύτο εταιριών. Πώς θα ε, παρεμποδίσουμε την αναστρατήγηση μέσω των σωστών ορισμών. Γιώτα Γιούτε Στάντο. Ε, πολύ γρήγορα πάτε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας. Άκουσα πολλά. Θέλω να μιλήσω λοιπόν έτσι απλά. Καταλήγω στο συμπέρασμα ότι χρειαζόμαστε μια κεντρική ευρωπαϊκή αρχή όπου να γίνονται έλεγχοι και επίσης να έρχεται και ενημέρωση γιατί έχω την εντύπωση όταν επιχειρήσουμε να τα επιλύσουμε όλα διμερός τότε υπάρχει τρομερή διοικητική επιβάρυνση. Μία κεντρική ευρωπαϊκή αρχή θα μας πήγαινε και, με, και συνδυασμένη με μία ευρωπαϊκή κοινωνική ταυτότητα για τους εργαζόμενους. Αν πάει κανείς εργοτάξια στη Γερμανία, για να ελέγξει τους εργαζόμενους, έχουμε το πρόβλημα ότι δεν είναι σαφής η κατάσταση όσον αφορά ποιος τους έχει αποστείλει, είναι πραγματικές εταιρείε ή είναι γραμματοκιβώτια. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάπου μια καταγραφή, ένας έλεγχος. Αλλά δεν το λέει η οδηγία αυτή. Αυτό. Τι θα κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις εταιρείες γραμματοκιβώτια. Πολύ συχνό πρόβλημα. Δεν θα τα σκόπιμο λοιπόν μια κεντρική αρχή να τα συντονίζει όλα αυτά. Μπορεί να τα λέω χοντρικά, αλλά ίσως θα μπορούσε να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε προς την επίλυση. Δεν βλέπω, λέει η Πρόεδρε, κανέναν άλλον. Να κάνω κι εγώ τις ερωτήσεις μου. Ήδη αναφέρθηκε σύντομα. Υπόθηκε ότι θα μπορούσαν τα επιτόπου συνδικάτα να εκπροσωπήσουν τους εργαζόμενους, αλλά καμιά φορά ούτε τα συνδικάτα επιτόπου, ούτε τα συνδικάτα της χώρας προέλευσης είναι σε θέση να εκπροσωπήσουν σωστά τους εργαζόμενους. Ποιος θα ήταν ο πιο κατάλληλος για να εκπροσωπήσει αυτούς τους εργαζόμενους, να τους δώσει στήριξη, πληροφόρηση, γιατί βρίσκονται σε μια ξένη χώρα. Τα συνδικάτα το κάνουν αυτό. Μήπως θα έπρεπε να είναι οι δημοτικές αρχές επιτόπου, μια κεντρική ευρωπαϊκή αρχή. Θα ήθελα να μάθω με βάση την πείρα σας. Α, παρακαλώ. Έχετε και σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Δεν ήθελα να υποβάλω ερώτηση γιατί με τους συμπειρογνώμονες ε, συνομίλησα πριν ε, τη συνάντηση, αλλά άλλαξα ιδέα τώρα. Στον κύριο Σλάιχερ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Μιλάμε για ορισμένα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι εταιρείε οι οποίες αποσπούν τους εργαζόμενούς τους. Εσείς ε, τι φρονείτε σχετικά με αυτή τη θεωρία που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα ανοιχτό κατάλογο, ένα κλειστό κατάλογο προϋποθέσεων που μπορεί όμως να είναι δύσκολο να τηρηθούν. Τι σκέφτεστε, παραλαμβάνω. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονές μας. Σας παρακαλώ να περιοριστείτε σε πέντε λεπτά. Καταλαβαίνω, είναι δύσκολο βέβαια σε πέντε λεπτά να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις που έχουν τεθεί, αλλά δυστυχώς ε, έχουμε λίγο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπύρ. Ελπίζω να μην το αφαιρέσατε και αυτό από το χρόνο μου. Ακούσαμε πολλές ερωτήσεις. Ο κύριος Κρίστενσεν, η κυρία Σρέτερ και η κυρία Τούρινεν αναφέρθηκαν ε, στους εργαζομένους που έχουν σύμβαση με γραφεία εξέβρεση προσωρινής απασχόλησης. Δημιουργείται μία θα έλεγα αμφίσιμη κατάσταση, διότι είναι δύο ε, οι εφαρμοστές οδηγίες. Είναι η οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων και η οδηγία για τα γραφεία εξέβρεση προσωρινής ε, απασχόλησης που εφαρμόζεται ταυτόχρονα. Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να διευκρινιστεί η κατάσταση. Ποιε είναι οι εφαρμοστέ ε, διατάξεις. Αν ε, κάνουμε μια διαπαραβολή των δύο οδηγιών, ε, καταλήγουμε στο προφανές συμπέρασμα πως οι πλανεκτικότερες συνθήκες εργασίας είναι εφαρμοστές για τους εργαζομένους μέσω είτε ή μάλλον θα πρέπει να έχουν τις πλεονεκτικότερες ε, συνθήκες εργασίας οι εργαζόμενοι, όποια και αν είναι η οδηγία που εφαρμόζεται. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας απλός ε, κανόνας. Ως προς ε, τον ορισμό του εργαζομένου, είναι μια ερώτηση που ακούσαμε πολλές φορές. Όπως είπε και ο κύριος Σλάιχερ, πριν από λίγα χρόνια έγινε διεξοδικότατη έρευνα για το θέμα των ψευδοαπασχολούμενων και γνήσιων αυτοαπασχολούμενων. Αυτό που μας εξέπληξε είναι ότι στο κατασκευαστικό τομέα χρησιμοποιείται ευρέως το σύστημα των ψευδοαπασχολούμενων για να καταστρατηγηθεί η εφαρμογή της οδηγίας περί Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα από του ελάχιστου ξεκάθαρου κανόνες σε σχέση με το τι εστί εργαζόμενο δεν υπάρχει ε, ε καταλαβαίνετε πόσο ε, αμήχανη κατάσταση για μα, διότι σε διεθνέ επίπεδο, σε επίπεδο διεθνού οργάνου εργασία υπάρχουν σαφέστατοι κανόνε. Αφήστε που ε, συχνά έχουμε νομολογία από πλευρά του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκή Ένωση για τα βασικά εφαρμοστέα κριτήρια, όμω δεν είναι υποχρεωτικά. Προτείνουμε λοιπόν ανεξαρτήτως από τη βούληση των ενδιαφερομένων, ε, να εξετάσουμε την ε, πραγματικότητα, την καθημερινή πραγματικότητα της εργασιακής σχέσης του εργοδότη και του εργαζομένου. Αν είναι γνήσια η αυτοαπασχόληση, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αν προκύψει όμως ότι ε, είναι ψευδής η εργασιακή σχέση, θα πρέπει να μετατραπεί σε κανονική σύμβαση απασχόλησης. Χρειαζόμαστε όμως κριτήρια. Το πρώτο είναι το κριτήριο της υπαγωγής subordination στα αγγλικά, όπως αναφέρεται στην πρόταση, θα πρέπει επακριβέστερα να ορίσουμε την έννοια του εργαζομένου. Αυτό με φέρνει σε ένα ιδιαίτερα λεπτό ζήτημα που ανέφερε η κυρία Τούρινεν. Τι συμβαίνει εάν δεν είναι εφαρμοστεία η οδηγία διότι υπάρχουν σετ κανόνων που εφαρμόζονται ταυτόχρονα, όπως σας έλεγα. Ακόμη και ε, οι νομομαθείς μας δεν έχουν ε, την ίδια άποψη σε σχέση με ε, αν είναι εφαρμοστεί η οδηγία της απόσπασης σε περίπτωση ψεύδου αν δεν υπάρχει πραγματική απόσπαση. Δηλαδή, είναι εφαρμοστέα η κείμενη εθνική νομοθεσία και οι συλλογικέ συμβάσει τη χώρα απασχόληση ή τη χώρα προέλευση. Αυτό δεν είναι ξεκάθαρο. Οι συζητήσει που γίνονται τώρα για την οδηγία περί εφαρμογής ε, είναι εξαιρετική στιγμή για να διευκρινίσουμε την κατάσταση. Για μας είναι προφανές όταν δεν υπάρχει σχέση απόσπασης, αλλά αποστέλλεται σε ένα άλλο κράτος ε, κάποιος εργαζόμενος, τότε είναι εφαρμοστεί οι κανόνες του κράτους ε, υποδοχής. Λαμβάνοντας επίσης ε, υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρχει ευνοϊκότερη μεταχείριση, για παράδειγμα, ευνοϊκότερη όρη αποζημίωσης της χώρας προέλευσης, που είναι ανύπαρκτη στη χώρα υποδοχής και αυτό θα πρέπει να συνυπολογιστεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα, διότι ε, αγγίζει ένα μεγάλο ρυθμό εργαζομένων που όμως δεν έχουν σχέση απόσπασης ε, με την ε, επιχείρησή τους. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα. Ποια συνδικάτα θα ήταν αρμόδια για να ασχοληθούν με το ζήτημα. Στις συζητήσεις που έχουμε κάνει στο ιστορικό των συνδικάτων για την ενημέρωση, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η οδηγία για τα εργασιακά συμβούλια, παραδείγματο χάρη, η οδηγία για την ευρωπαϊκή εταιρεία. Υπάρχουν νομοθετικές διατάξεις για την ενημέρωση. Παραδόξως όμως στους ε, πολυεθνικούς χώρους εργασίας, όταν εργάζονται στον ίδιο χώρο ε, με υπήκοοι διαφόρων χωρών, ε, υπάρχει κενό στην νομοθεσία. Αν εξετάσουμε την νομοθεσία και δεν εφευρίσκουμε εδώ κάτι καινούριο, συνειδητοποιούμε ότι μπορούμε για τη διαβούλευση και για την ενημέρωση να χρησιμοποιήσουμε τις ίδιες διατάξεις ακόμη και για αυτούς τους ε, διεθνικούς ε, χώρους εργασίας. Ε, σε μια πρόσφατη υπόθεση στην Ολλανδία και θα σας συμβούλευα να διαβάσετε τη σχετική, το σχετικό έγγραφο. Ε, ε, υπάρχει ένας παρόμοιος μηχανισμός. Έχουμε ακόμη και συλλογικές συμβάσεις. 500 ε, Πολωνοί μισθωτοί είχαν σημαντικότατη αύξηση μισθού χάρη σε αυτό το μηχανισμό για την προσκόμιση πληροφοριών. Όλα τα συνδικάτα θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους χώρους εργασίας, ε, επιτελώντας έτσι αυτό το ρόλο ενημέρωσης. Θα αφήσω τώρα το λόγο στους ε, ε, συναδέλφους για να μην απαντήσω εγώ όλες τις ερωτήσεις, δεν θα ήταν ευγενέ εκ μέρους μου. Σας ευχαριστούμε. Ας ακούσουμε τώρα τον καθηγητή Γιόρενς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, δεν είμαι σίγουρος ότι θα απαντήσω σε, στις υπόλοιπες ερωτήσεις, γιατί μπορεί να έχω διαφορετική απάντηση στις ήδη απαντηθήσεις ερωτήσεις. Σίγουρα δεν προλαβαίνω να τα πω όλα αυτά που θέλω να πω σε πέντε λεπτά. Ποιο, τι θεστεί αποσπασμένος εργαζόμενος, σε ποιο συνορισμός και ποιον καλύπτει. Νομίζω ότι η πρόταση περί εφαρμογής ε, αξίζει εύσημα διότι προσδιορίζει τα κριτήρια και τον ορισμό αυτών των εργαζομένων ε, διότι η Οδηγία γεννά πολλά ερωτηματικά. Ποια είναι η εφαρμοστέα νομοθεσία, αναρωτιόμαστε. Μα είναι ο κανονισμό Ρώμη 1, που είναι το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να δούμε προς τα που κατευθυνόμαστε, διότι υπάρχει η μητρική αυτή η νομοθεσία, στη χαρακτηρίσω έτσι, σε σχέση με το θέμα της απόσπασης και άρα θα πρέπει να εξετάσουμε όλες τις διατάξεις και τους κανόνες του κανονισμού Ρώμη 1 για να ε, διαπιστώσουμε ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο σε ποια περίπτωση. Η ψευδοαυτοαπασχόληση αναφέρθηκε επανειλημμένα ε, στη συζήτησή μας. Μάλιστα, είναι ένα από τα πιο καυτά ζητήματα. Το πρόβλημα εδώ σχετίζεται με το θέμα ε, της αρμοδιότητας. Μπορείτε να ισχυριστείτε ό,τι θέλετε για το, την ευρωπαϊκή διάσταση. Ε, έχει κάνει κάποιες υποδείξεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έμεσα παραπέμπει πάντοτε στην εθνική νομοθεσία ε, για να στοιχειοθετηθεί ε, ποιος είναι γνήσιος ή ψευδός αυτοαποσχολούμενος. Σε τώρα με την θέσπιση ευρωπαϊκών κριτηρίων για το ζήτημα αυτό ενδέχεται να προκύψει σοβαρή σύγκρουση ανάμεσα στην εθνική και αρμοδιότητα και την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να να αναγνωρίσουμε ότι θα υπάρξει διάσταση απόψεων σε σχέση με ε, το τι υπερισχύει, ποια νομοθεσία υπερισχύει. Για τις ε, διάφορες οδηγίες, τώρα η οδηγία για τα γραφεία εξέβρεση προσωρινής απασχόλησης ε, κτλ. Κοιτάξτε, είναι ένα είδος ε, αυτοαπασχολούμενων όσοι έχουν σύμβαση με τέτοια γραφεία, αλλά καλό θα ήταν πάντως να ληφθεί αυτό υπόψη από όσους εξετάσουν αυτές τις δύο οδηγίες. μιλήσατε για μια ευρωπαϊκή μέθοδο επίλυσης των προβλημάτων, σαν ονείροξη μου ακούγεται. Ε, το πρόβλημα έγκυται στην έλλειψη ε, συνεργασίας ανάμεσα στις ε, αρχές αρμόδιες για την επιθεώρηση. Η μαύρη εργασία στη Γερμανία ελέγχεται από μια διοικητική υπηρεσία. Ε, στην Αυστρία είναι φορολογική υπηρεσία. Ε, αυτή η σοσιοπόλη, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Αστυνομία για θέματα κοινωνικά τέτοια, είναι ένα δύσκολο ζήτημα διότι ε, τίθεται αυτό το ζήτημα αρμοδιοτήτων εγώ πάντως είμαι σαφέστατα υπέρ και θα σταματήσω ε, στα τέσσερα λεπτά. <laughs> Thank you. Uh, Σας ευχαριστώ και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Νόγκαρντ. Ευχαριστώ. Ε, προς τον κύριο Κρίστενσεν γιατί το θέμα των μεταφορών, ναι, όντως είναι δύσκολο το ζήτημα και στη Δανία προς το παρόν αναλύουμε την κατάσταση για να καταλάβουμε πώς στον τομέα των μεταφορών μπορούμε να επιτύχουμε ορθότερη εφαρμογή. Μιλάμε για το καμποτάζ, όπου εφαρμόζεται η οδηγία για την απόσπαση. Όμως υπάρχουν προκλήσεις διότι είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος απασχόλησης και υπάρχουν και διαφορετικοί χώροι εργασίας. Ε, το καμποτάζ έχει ειδικό του κανόνες, έχουμε τους εθνικούς κανόνες, έχουμε και τις συνδυασμένες μεταφορές, άλλο ξεχωριστό κεφάλαιο πάλι. Αν ε, προκύψουν καλές ιδέες ε, θα σας τις διαβιβάσουμε. Σχετικά με το A1, Α1, αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ε, όργανο ελέγχου. Οι εργαζόμενοι μπορούν να το επικαλεστούν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες περιπτώσεις όταν αποστέλλεται το εργαζόμενος σε κάποια άλλη χώρα αρκεί να αποδειχθεί ότι υπάρχει ουσιαστική επαγγελματική δραστηριότητα στην χώρα προέλευσης. Όμως ε, θα πρέπει να θεσπιστούν κάποια αντικειμενικά τεκμήρια σχετικά με το αν ναι, ε, μπορεί να επικαλεστεί αυτή τη διάταξη ο Εάν τώρα θέλετε να θεσπίσετε σύστημα κοινή ευθύνη, είναι μάλλον πολιτικό το ζήτημα. Η κυρία Σρέντερ όντως με παρανόησε. Στο τέλος ανέφερα ότι ε, αποτελεί καλό εφαλτήριο η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όμως ε, μιλώντας για το άρθρο 9 παρά ήμουν ε, διπλωμάτης. Ο κύριος Σλάιγερ ήταν πολύ πιο όμως και άμεσος. Μπορώ όμως να προσυπογράψω τη θέση του, είναι και η θέση της Δανίας εξάλλου. τι πρέπει να κάνουμε, λένε κάποιοι να διαγράψουμε το άρθρο 9 ή να περιορίσουμε τη χρήση του, να βρούμε τη μέση λύση. ανάμεσα στην κατάργηση και την περιορισμένη χρήση. Εμείς αυτό εξετάζουμε αυτή τη στιγμή. Κυρία Τούρινεν, για τους ορισμούς. Η οδηγία των 96 που υποτίθεται μας δίνει τον ε, ορισμό του εργαζομένου στη χώρα υποδοχής ε, έχει ως αποτέλεσμα να έχετε την εργασιακή σας σύμβαση στη χώρα προέλευσης και παρόλα αυτά να εργάζεστε στη χώρα ε, υποδοχής, αλλά περιπλέκονται τα πράγματα όταν αποκτά ε, ε, διασυνοριακή διάσταση ε, το πράγμα. Σε σχέση τώρα με τον κανονισμό Ρώμη 1, αυτή τη στιγμή αναλύουμε τις επιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 3 σε περιπτώσεις όπου κάποιος δεν καλύπτεται από την οδηγία περί απόσπασης. Σημαίνει αυτό ότι η χώρα υποδοχής μπορεί να εφαρμόσει την ε, κείμενη νομοθεσία ή την οδηγία Ρώμη 1, γιατί αυτό συνεπάγεται ότι μια εντελώς διαφορετική χώρα από τις δύο εμπλεκόμενες ε, ε, μπορεί να, ενδέχεται να έχει την αρμοδιότητα για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Για το κεντρικό αυτό σύστημα, όπως σας είπα, εδώ και καιρό επιθυμούμε την θέσπιση ενός τέτοιου συστήματος, αλλά θα είναι δύσκολο να υλοποιηθεί το πρόγραμμα γιατί ακόμη και η Δανία θα πει είναι καλή ιδέα αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη, την τάδε ή τη δίνα παραχώρηση, αυτό είναι εθνικό ζήτημα και ούτω καθεξής. Είναι μεγάλη ε, πρόκληση δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος αλλά ε, πάντοτε τετοιου συστηματος αλλα μπορεί να έχει τις φιλοδοξίες του. Ως προς τις εικονικές επιχειρήσεις, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα και στην Δανία είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαπιστώσουμε αν είναι εγκατεστημένη, έχει την έδρα τη μια επιχείρηση στη Δανία, αλλά δραστηριοποιείται και σε άλλε χώρε, ε, είναι δύσκολο να διαπιστωθεί αν ε, είναι πραγματική εικονική. Ε, η πρόταση πάντως για την εφαρμογή της οδηγίας όντως περιέχει μηχανισμούς που θα διευκολύνουν την εφαρμογή και θα διευρύνουν την εφαρμογή της οδηγίας σε περισσότερες περιπτώσεις. Thank you. And now Mr. Schleicher, please. Ο κύριος Schleicher. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει πολύ ε, χρόνος, οπότε θα μιλήσω γερμανικά. Α, μάλιστα, ωραία. Τονίζω λοιπόν Είμαι επιχειρηματία στον τομέα των ε, κατασκευών, όχι διπλωμάτης. Οπότε ορισμένα τα λέω στα Ωστόσο είμαι και πρόεδρος της ΦΙΕΚ. E Για πολλές άλλες λοιπόν κατασκευαστικές εταιρείες επίσης μιλάω. Πρώτον, τι μπορεί να κάνει κανείς. για να βελτιώσει την ανταλλαγή πληροφοριών. Θα πρότεινα να κοιτάξετε το κοινό website που έχει η εταιρεία των εργαζομένων, η εταιρεία των εργαζομένων στον τομέα των κατασκευών και η Ομοσπονδία των Εργοδοτών. Εκεί μπορούν να δουν τα δικαιώματά τους σε κάθε μια χώρα υπάρχει πληροφόρηση από ε, τις, τους κοινωνικούς εταίρους, από τα Υπουργεία εργασία ή τις άλλες διοικητικές αρχές των κατά χωρών. Οι χώρες, αν θέλουν, μπορούν να εισαγάγουν πληροφόρηση. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. και με αυτόν τον τρόπο μπορεί οποιοδήποτε αποστέλλεται κάπου και η, η εταιρεία που τον αποστέλλει να ξέρει τι τον περιμένει στη χώρα υποδοχή. Δεύτερον, η πρόταση να υπάρχει μια κεντρική υπηρεσία. Το ερώτημα αν είναι σκόπιμο να κάνουμε μια τέτοια κεντρική υπηρεσία για να βελτιώσουμε την κατάσταση της ενημέρωσης δεν μας βρίσκει συμφώνους. Δημιουργούμε τεράστια γραφειοκρατία και υποθέτω ότι η ενημέρωση μέχρι να φτάσει σε αυτή την ε, κεντρική υπηρεσία θα είναι ήδη ξεπερασμένη. Όχι λοιπόν, καμία κεντρική αρχή. Και δεν νομίζω ότι είναι θέμα της Ένωσης να φτιάξει μια κεντρική λύση για όλα τα προβλήματα σε όλες τις χώρες για τα θέματα των εργαζομένων που αποσπώνται. Υπάρχουν πολλά θέματα διμερών σχέσεων στην Ευρώπη οι διμερείς σχέσεις για παράδειγμα μεταξύ Γαλλίας και Πολωνίας, μεταξύ Ισπανίας και Πολωνίας και Γερμανίας και Πολωνίας είναι διαφορετικές. Και επειδή πάκτα σουν σερβάντα έχουν οδηγήσει ή κάθε φορά διμερείς αυτές σχέσεις τα βέλτιστα αποτελέσματα. Δεν νομίζω ότι θα μα βοηθούσε στην Ευρώπη η συνεχής προσπάθεια υπερσυγκεντρωποίησης οι συμβάσεις με τις νέες χώρες της ε, Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι διαφορετικές και για λόγους γλωσσικούς ε, με τις συμβάσεις που υπάρχουν μεταξύ χωρών που ήταν ήδη από παλιά χώρες της Ένωσης. Πώς μπορούμε να επιτύχουμε την βελτίωση της ροής ενημέρωσης σε κάθε χώρα μόνο μέσω ισομερού συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Υπάρχει μια οργάνωση εδώ στι που λέγεται AIP, που ασχολείται με την εργασία όλων των ισομερών ε, οργανώσεων. Είναι πολύ επιτυχή στη δράση τη. Ω επιχειρηματία, μπορώ να σα πω ότι εμεί στη Γερμανία, για παράδειγμα, έχουμε το σύστημα ενημέρωσή μα όσον αφορά αποσπόμενους εργαζομένους ε, είναι τόσο τελειοποιημένο ούτω ώστε να μην τίθεται καν το θέμα πλέον ε, εταιριών γραμματοκιβωτίων. Μαζί λοιπόν με τους κοινωνικούς εταίρους και ε, το κοινωνικό ταμείο λειτουργεί έτσι το σύστημά μας, ούτω ώστε κανείς δεν προσλαμβάνει ανθρώπους από τέτοιου είδους ε, ψευδοεταιρείες. Ξέρετε ότι κανείς δεν κάνει εκ προθέσεως ε, τέτοιου τύπου αδικήματα, αλλά ξέρετε ότι ε, στις διαπρα... συλλογικές διαπραγματεύσεις προσπαθούμε να αποφύγουμε αυτά τα φαινόμενα. Τελευταία ερώτηση. Ποιος εκπροσωπεί τους εργαζόμενους... Α, κάτι άλλο, για το άρθρο 9. Νομίζω ότι το περιεχόμενο του άρθρου 9, οι δυνατότητες ελέγχου που κάποια κράτη-μέλη ικανά έχουν ήδη, την περιορίζουν. Οπότε, όπως έχει τώρα, το άρθρο 9 το απορρίπτω. Δεν νομίζω ότι είναι επαρκές. Ποιο εκπροσωπεί τους εργαζόμενους, ε, τους αποσπασμένου στη χώρα υποδοχή, Αυτό είναι πρόβλημα των συνδικάτων, όχι τη διοίκηση. Για μας, όταν υπάρχουν διαφωνίε που δεν μπορούν να επιληθούν ε, μέσω μιας οδηγίας, τότε ισχύει το εθνικό δίκαιο τη χώρα υποδοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σλάχια. Τέλος, να ξαναδώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας, Τανούτα Κλατσοβιέτσκα. Ζητώ συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Δεν άκουσα κανένα να απαντάει στη δική μου την ερώτηση. Παρακαλώ τον κύριο Σλάιχερ, τι ακριβώς σκέφτεται για τα κριτήρια που θα πρέπει να σέβονται οι εταιρείε σχέτιση με την οδηγία. Ναι, με συγχωρείτε. Τα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται καθορίζονται στο άρθρο 9. Νομίζω ότι σε διάφορες χώρες ήδη υπάρχουν πολύ ευρύτερα κριτήρια πιο πολύ άριθμα. Οπότε τα αναφερόμενα κριτήρια και οι περιορισμοί μου επαρκούν. όχι, δεν μου επαρκούν. Είναι, πιστεύω ότι δεν είναι επαρκή αυτά που ζητούνται στο άρθρο 9. Ξέρω ότι υπάρχουν χώρες που τα κριτήρια που καθορίζονται τώρα στο άρθρο 9 είναι τέρα incognita για σε άλλες χώρες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εμπειρογνώμονές μας, οι οποίοι ήταν πλήρως προετοιμασμένοι. Τους ευχαριστώ για τις εισηγήσεις τους. Συνάδελφοι, εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ασχολούμαι με αυτή την οδηγία. Δεν ξέρω εάν το ασυμβίβαστο μπορώ να το συμβίβασω, ε, αλλά τουλάχιστον εύχομαι ελπίζω να μπορέσω να συντάξω ένα κείμενο που να καλύπτει και τους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Αλλά το έργο αυτό δεν θα είναι δύσκολο, δεν θα είναι εύκολο συγγνώμη. Γιατί μιλάμε για αποσπασμένους εργαζόμενους που εγκαταλείπουν ένα κράτο μέλος και πάνε σε ένα άλλο. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ένας μέσος πολίτης, αν δεν αντιμετωπίζει δεινά προβλήματα, ε, όταν πηγαίνει σε μια άλλη χώρα δεν αντιμετωπίζει τις ίδιες συνθήκες κατά τις οποίες θα εργαζόταν στη δική του τη χώρα. Να υπενθυμίσω ότι οι διάφορες χώρες ε, είναι εντελώ διαφορετικές μεταξύ τους. Είναι λοιπόν δύσκολο να τα συνδυάσουμε όλα αυτά αλλά είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι από τα βασικά σημεία που μας απασχολούν. Επίσης, θα πρέπει να συλλογιστούμε και το, ας το πούμε, τον ξεριζωμό αυτών των εργαζομένων που πηγαίνουν σε ένα άλλο κρότος Μία από τις αδυναμίες της οδηγίας είναι η έλλειψη ενημέρωσης πληροφοριών αξιόπιστων, ενημερωμένων και να υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες στη διάθεση των αποσπαζόμενων και δεν υπάρχει επικοινωνία μάλλον καλύτερα να το πω, όχι περισσότερο από ότι όχι πλήρω ενημέρωση. Αυτό είναι το πραγματικό, το βασικό πρόβλημα. Είναι το κουτί της Πανδώρας. Και τελικά όταν μιλάμε ότι, και λέμε ότι δεν υπάρχει πληροφορία, τότε να η απάτη, να τη συμβαίνει. Δεν υπάρχει μια, ένα συντονισμός ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα κράτη-μέλη θα καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να προστατεύσουν καλύτερα και τους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Από τα εργαλεία που μπορούν να το πετύχουν αυτό είναι το σύστημα ενημέρωσης ανακοίνωσης ε, ε αναλύσαμε τις συστάσεις ε, των ε, εισηγητών μας. Σε 18 κράτη-μέλη έχουμε παρόμοια συστήματα ενημέρωσης που διαφέρουν όμως το ένα από το άλλο. Και ανάμεσα στους εργοδότες υπάρχει ένα κομφούζιο μπορούμε να πούμε. Δεν ξέρουν ακριβώς ο καθένας τι γίνεται. Χρειάζεται να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων και δεν λύνεται και το πρόβλημα των ελέγχων που έθιξαν οι συγκεκριτές μας. Ο καθηγητής κύριος ε, Γιώργος μας είπε ότι η ενιαία αγορά δεν προσφέρει και ίσες δυνατότητες. Θα πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί, αλλά θα πρέπει να είμαστε και φιλόδοξοι για να συντάξουμε ένα κείμενο, για να ε, αφαιρέσουμε αυτές τις προϋποθέσεις ε, τις απαραίτητες για τις ψευδοεπιστήμες. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Ε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσε οι παρεμβάσει σα. Καλό ταξίδι, καλή επιστροφή. Και τέλος Νοεμβρίου θα συζητήσουμε την ε, έκθεση και τροπολογίες μέχρι 13 Δεκεμβρίου 12 το μεσημέρι. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα της μέρης διάταξης. Um, so kind, Ever so Okay. Um, Herr Händel, wir haben ein kleines... Κύριε Händel, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Θα συμφωνούσατε να κάνουμε μία εναλλαγή μεταξύ της δικής έκθεσης και της έκθεσης Μακεντάερ. Ο κύριος Χέντελ, σε τρία τέταρτα πρέπει να μιλήσω αλλού για τις συμβάσεις παραχώρησης, αλλά εντάξει. Εντάξει, ωραία. the noise, because otherwise it's impossible. Ich würde ich würde die Leute I would like ask you to leave. Παρακαλώ φεύγοντας μην κάνετε πολύ θόρυβο. Εν πάση προχωράμε. Λοιπόν, παρακαλώ Περνάμε στο θέμα 26. Έκθεση McIntyre. Πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δυνατότητες χρηματοδότησης. Θα δώσω λόγο στην κυρία McIntyre. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που επιτρέψατε να συζητήσουμε τώρα το θέμα αυτό. Προσπάθησα να κανονίσω πριν από την εκθεσή μου μια συνεδρίαση των σκιωδών. Δεν κατέστη δυνατόν. Αλλά χαίρομαι που χαλάρωσα αρκετά το χρονοδιάγραμμα εξέταση αυτή τη έκθεση. Θα έχουμε λοιπόν πολύ περισσότερο χρόνο για να υποβληθούν τροπολογίες για να το συζητήσουμε για συνεδριάσεις των σκιωδών και τροπολογίες αντί απλώς να υποβληθούν στα αγγλικά μπορούν να υποβληθούν σε όλες τις γλώσσες. Χαίρομαι πολύ που η ΕΚΟΝ παρέτεινε τις προθεσμίες για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε σκοπιμότερα. Ελπίζω να συνεχιστεί το θαυμάσιο επίπεδο συνεργασίας που είχαμε στην προηγούμενη γνωμοδότηση που έκανα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το περιεχόμενο τώρα. Ξέρουμε ότι οι γνωμοδοτήσεις ε, έχουν περιορισμένο μήκος. Υποθέτω λοιπόν ότι θα υποβάλω και εγώ κάποιες τροπολογίες και ορίζω και τις ενδεχόμενες ε, τροπολογίες των συναδέλφων. Προσπάθησα να μην ξανακάνουμε την εργασία της επί της ουσίας επιτροπής, αλλά να περιοριστώ στις πλευρές απασχόλησης. Κάποια θέματα σύντομα. Ως Επιτροπή διαπιστώσαμε και προηγουμένως ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, απασχολούν 90 εκατομμύρια εργαζόμενων και 85% των νέων θέσεων εργασία δημιουργούνται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσει. Η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει τους επιχειρηματίες και τις μικρομεσαίες πάρα πολύ έντονα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βεβαίως υποφέρουν, οπότε μειώνονται και οι, δημιουργοί, και οι νέες θέσεις εργασίας. Σημειώνουμε ότι το επιχειρηματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται μόνο από 7% των ΜΜΕ και 60% των επιχειρήσεων λένε ότι το επιχειρηματικό κεφάλαιο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιχείρησή τους. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε άλλες πρωτοβουλίες, όχι τραπεζικοί όπως ε, μικροδανισμούς, από επιχείρηση σε επιχείρηση και ελπίζω η Επιτροπή να το στηρίξει αυτό. Για να δείτε πόσο επίκαιρο είναι το θέμα αυτό και σημαντικό, στη χώρα μου είδα μια έκθεση όπου λέγεται ότι δύο τρίτα των επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν θεωρούν ότι είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητες ε, χρηματοδότησης και πολύ λίγες επιχειρήσεις ε, θεωρούν ότι είναι η όρη χρηματοδότησης ε, λογική. Θέλουμε λοιπόν να συνεργαστούμε με τους κοιόδης και θα ακούσω ε, με πολύ ενδιαφέρον τα σχόλιά τους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Θέρκας. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ. Κύριε Μακιντάιρ, ναι, εδώ, εδώ, εδώ είμαι μπροστά σα, απέναντί σα, μάλλον. Αντικαθιστώ την κυρία Ράπτη που θα αργάστηκε να αναχωρήσει για την Ελλάδα. Ξέρετε ότι με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουμε πολλά προβλήματα στην Ελλάδα και τώρα στην Αθήνα λαμβάνει η χώρα μια συνάντηση, έπρεπε να παραστεί και μου ζήτησε να σας πω μερικά πράγματα βασικά ουσιαστικά για τους σοσιαλιστές. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εργασία σας και να σας πω ότι σίγουρα θα συνεργαστούμε. Το είπατε, δεν είναι μόνο οικονομικό το πρόβλημα, αλλά πάνω απ' όλα ότι ίσως ε, είναι εκεί που οφείλονται όλα τα δεινά μας ε, σε πάρα πολλές χώρες ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ακριβώς το 90% του συνόλου της απασχόλησης και πολλές χώρες μας το 90% τους απασχόλησης που χάθηκε είναι ότι αυτές εξαφανίστηκαν, αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το 90% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εξαφανίζονται στις χώρες μας, τουλάχιστον στη Ισπανία, στη δικιά μου χώρα, ε, πέρα από το ειδικό πρόβλημα ακριβώ της φούσκας της ε, οικοδομικής είναι επειδή δεν πετυχαίνουν χρηματοδότηση. Για αυτό δεν έχουν από πού να πάρουν χρήματα. Δεν χρηματοδοτούνται. Γι' αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να μιλήσουμε για την προοπτική αυτή της απασχόλησης και θα ήθελα επίσης να σας πω ότι θα υποβάλουμε, θα καταθέσουμε μια τροπολογία ε, για δύο συγκεκριμένα σημεία. Πρώτα απ' όλα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι τα εργαλεία, τα μέσα. Αλλά λείπει, λείπει τρομερά η ενημέρωση και δεν χρησιμοποιούνται μερικές φορές αυτά τα εργαλεία γιατί δεν ξέρει κανείς, δεν το ξέρουν ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τι αξίζει τώρα να υπάρχουν προγράμματα και μέσα αν οι τελικοί λήπτες δεν τα γνωρίζουν έτσι και μάλιστα εκείνοι που είναι περισσότερο στο, περιθώριο είναι πιο απομακρυσμένοι. Και το δεύτερο που θέλαμε να σας πούμε είναι ότι τώρα, κυρίως σε χώρες του νότου της Ευρώπης, όπου μειώνεται η ζήτηση όλες οι επιχείρησεις, ε, η ελπίδα τους είναι να πάνε σε εξωτερικές αγορές ε, και γι' αυτό η διάσταση αυτών των ε, οικονομικών ενεργειών και πάντα υπέρξαν προβλήματα εκεί πολύ μεγάλα και δεν υπάρχει χρηματοδότηση βέβαια τώρα για να μπορέσει κανείς να αντιμετωπίσει αυτό που είναι το όνειρο που δεν μπορούν να πετύχουν, να πάνε σε άλλες αγορές και εκεί να βρουν τη ζήτηση που δεν βρίσκουν στην αγορά τους. Αυτά λοιπόν η διεθνοποίηση αυτών των οικονομικών δραστηριοτήτων και την υποστήριξη για να μπορέσουν να βγουν σε άλλες αγορές αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λοιπόν, θα πρέπει να είναι κάτι που χρειάζεται ρητά και κατεγραμματικά να αναφέρει, να θίγει η έκθεσή σας. Επιθυμείτε και πάλι το λόγο. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, να απαντήσω σύντομα. Ευχαριστώ πολύ επικοδομητικά σχόλια. Έλλειψη ενημέρωση, είπατε. Ελπίζω το σημείο 7 ε, να αντιμετωπίζει κάπως το θέμα όπου μιλάμε για την έλλειψη γνώσης και ενημέρωσης που μπορεί να θίξει την παροχή κτλ. Και η ανάπτυξη των εξωτερικών αγορών. Συμφωνώ. Αν αυτό αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, αυτό το είπαμε στην προηγούμενη γνωμοδότησή μας για τις ΜΜΕ. Πώς πρέπει να τις βοηθήσουμε να εξαγάγουν. Φυσικά θα λάβω υπόψη και θα συμπεριλάβω οποιασδήποτε τροπολογίες που βάλετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Όπως υπόθηκε, η ΕΚΟΝ ανέβαλε την ψηφοφορία της, οπότε για μας η τροπολογία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι 2 Οκτωβρίου, η προθεσμία υποβολή τροπολογιών και ενδεχομένω 6 Νοεμβρίου να συζητήσουμε τις τροπολογίες αλλά τότε θα πρέπει να κάνουμε μια επιπλέον συνεδρίαση. Δεν είναι λοιπόν σίγουρη αυτή η ημερομηνία ακόμη. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 29 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε πηδάμε τώρα στο 25 πάλι πίσω, επανερχόμεθα στην ε, ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης και το λόγο έχει ο συγητής κ. Χέντελερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να δώσουμε γνωμοδότηση στην ΙΜΚΟ για το θέμα συμβάσης παραχώρησης. Πρόκειται για μια νέα οδηγία που δεν υπάρχει προηγούμενο. Είναι λοιπόν ε, νέο έδαφος εδώ. Αυτή η οδηγία αυτή συζητήθηκε ήδη προκατακτικά στην έκθεση Ρούλε το 2011. Το Κοινοβούλιο είχε τότε σημαντικές αμφιβολίες αν θα έπρεπε να γίνει οδηγία ή όχι. Αμφιβάλλουν και πολλοί εμπειρογνώμονες γι' αυτό που εκφράστηκαν στα πλαίσια της προκαταρκτικής συζήτησης. Και άλλες αφιβολίες αφορούν την περιπλοκότητα του αντικειμένου που είναι τόσο περίπου και οι δημόσιες προμήθειες. Δεν θέλουμε λοιπόν να προκύψει μια κατάσταση του χρόνου λοιπόν να χρειαζόμαστε μια σειρά από μεταβατικές ε, οδηγίες για να μπορέσει επιτέλους να εφαρμοστεί αυτό που θα αποφασίσουμε τώρα σε πολλές χώρες και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο έθεσε θέμα επικουρικότητας και είπε ότι θα κάνει προσφυγή. Υπάρχουν λοιπόν αμφιβολίες. Την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να το συζητήσουμε με τον εισηγητή Ίμκο. Η Ίμκο μέσω του εισηγητή αποφάσισε να ζητήσει μια εντελώς νέα εκδοχή για την οδηγία αυτή, αλλά αυτό δεν απλοποιεί την κατάσταση. Σε ένα σημείο υπάρχει αρκετή ομοφωνία και αυτό προκύπτει και από τις τροπολογίες. Φοβούνται ορισμένοι ότι θα ε, κατά πολύ η δυνατότητα δράσης διαφόρων δημοσίων αρχών και επίση, φοβούνται ότι θα υπάρξουν διαφωνίε για τις ε, αρμοδιότητε των ΜΕΝ και των ΔΕΛ και για την παροχή λοιπόν σημαντικών υπηρεσιών ε, κοινή ωφέλεια. Έχουμε 80 τροπολογίε. Πολλέ ασχολούνται με τα ίδια θέματα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους Εστρέλα, Τσουλιμάνε και Μανέσκου γιατί νομίζω ότι οι τροπολογίε του πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Θα επιχειρήσουμε να συναντηθούμε, να συμφωνήσουμε για τις ήδη διατυπωθήσεις συμβαστικέ προτάσει. Θα αναφέρω μερικά σημεία τώρα πολύ σύντομα. Η οδηγία αυτή λέει στην αρχή ότι αν πρόκειται να γίνουν συμβάσει παραχώρηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι απλώς ε, η φθηνότερη τιμή, αλλά η οικονομικά πιο συμφέρουσα πρόταση. Ε, βεβαίως υπάρχει μια τροπολογία που επιδιώκει να ξαναβάλει την ε, ιδέα της υπηρεσίας σε σχέση με την τιμή αυτή τροπολογία 48 με, από την πίσω πόρτα λοιπόν προσπαθεί να επανέλθει το κριτήριο μόνο τη τιμή. Θέλουμε να το απορρίψουμε. Δεύτερο το θέμα ε, προστασία των ε, συνδικών εργασία, ε, δηλαδή συλλογικέ συμβάσει βεβαίω και σύγκριση των αποδοχών για την ίδια εργασία στον ίδιο τόπο. Τρίτο σημείο, το θέμα όταν ε, η μία, παραχώρη, η μία παραχώρηση πηγαίνει από μία εταιρεία στην άλλη, πρέπει να υπάρχει μία μεταβατική περίοδος και διατάξεις γι' αυτό. έχει να κάνει και με αυτό που είπαμε προηγουμένω Όχι το θέμα της ευθύνη σε αλυσίδα, αλλά ποιο έχει την τελική ευθύνη. Επίσης, το θέμα της ε, διαφάνειας νομίζω ότι θα έχουμε συμφωνία. Χαιρετίζω ιδιαίτερα το ότι η Κομισιόν στην πρότασή της το τομέα εκπαίδευση κοινωνικών υπηρεσιών και ε, υγεία τους έχει εξαιρέσει τους τομεί αυτού. Θα πρέπει επίσης να δούμε και τις υπηρεσίες στον τομέα του πολιτισμού, το, της αποχέτευσης, των απορριμμάτων και της ίδρυυσης. Αυτά τα θέματα θα τα δούμε όταν θα συζητήσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες. Σημαντικό είναι αυτό που αναφέρουν συνάδελφοι σε κάποιες ε, τροπολογίες, το να μην υπάρχουν διακρίσεις και το θέμα της ισότητας των φύλων. Νομίζω ότι για τα θέματα αυτά μπορούμε να συμφωνήσουμε. Υπάρχουν τιμία, σημεία τομή. Για τι άλλε τροπολογίε θα κάνω τις αντίστοιχε προτάσει. Και θα επιδιώξω μέσω τη συζήτηση να καταλήξω σε πλειοψηφία ε, στην Επιτροπή μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή πρώτα απ' όλα σχετικά με τις σημαστικές τροπολογίες που μας έστειλε. Να τον συγχαρώ για την εξαιρετική εργασία του. Μετά από μία πρώτη ανάλυση, κρίνω ότι η πολιτική μου ομάδα θα μπορέσει να υποστηρίξει αυτές τις σημαστικές τροπολογίες, διότι θεωρώ πως ναι, υπάρχει κάποιο θέμα με τη διερμηνία, δεν ακούτε. Ξαφνικά ακούω δανέζικα στα ακουστικά μου, λέει ο εισηγητής. It's okay. Ich hoffe. It's okay now. <laughs>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 Λοιπόν, θα επαναλάβω αυτά που έλεγα. Σας χάρη για την εργασία σα. Σα ευχαριστούσα για τι συμβαστικές τροπολογίε που μα στείλατε. Μετά από μία προκατακτική ανάλυση θεωρώ ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ώστε η πολιτική μου ομάδα να υποστηρίξει αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες στο βαθμό που καλύπτονται και οι δικές μου τροπολογίες μέσω των συμβαστικών τροπολογιών και ανταποκρίνονται στο στόχο μας. Όντω, ε, επιφέρατε βελτιώσεις σημαντικές στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έξω ε, και τα συγχαρητήρια για το έργο σας. Προσπαθείτε να καλύψετε τις ανησυχίες ε, των ε, εταίρων που ανησυχούσαν για τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της οδηγίας αυτής ε, στην καθημερινή δουλειά τους. Εισαγάγονται τώρα κοινωνικά κριτήρια για την ανάθεση παραχωρήσεων. Υπάρχει το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής, όπως σωστά αναφέρατε κι εσείς, αποφεύγοντας έτσι περιπτώσεις κοινωνικού ντάμπινγκ. Υπέβαλα διάφορες ε, τροπολογίες, ε, πάνω κάτω 25, με στόχο την αυξημένη διαφάνεια για τα κριτήρια που διέπουν αυτές τις συμβάσεις παραχώρης, αποφεύγοντας έτσι στρεβλώς στην εσωτερική αγορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατοχυρωθούν αυτά τα κριτήρια κοινωνικού περιεχομένου και οι βασικές διεθνείς συμβάσεις για κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα επίσης πρέπει να γίνουν σεβαστές στη διαδικασία ανάθεσης παραχωρήσεων. συνοπτικά θα έλεγα ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε την προεξάρουσα θέση των οικονομικών κριτηρίων σε αυτές τις συμβάσεις για να χρησιμοποιηθούν και άλλα κριτήρια βιωσιμότητας, περιβαλλοντικά κριτήρια, κριτήρια πρόσβασιμότητας ε, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες κτλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να θέλει κανείς άλλο το λόγο. Κύριε Χέντελ, θέλετε να πείτε τίποτα περαιτέρω. Όχι, λόγω και του χρόνου. Έγινε λοιπόν η πρώτη ανταλλαγή. Σε 20 λεπτά θα επιχειρήσουμε να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε επί των συμβαστικών προτάσεων. Δεν βλέπω να υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μια ανακοίνωση από τη συνάδελφο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Συντομότατη θα είμαι όπως είπε συνάλφος Χέντελ που τον ε, συγχαίρω είναι πολύ τεχνικής φύσεως και πολλά δεν εμφανίστηκαν ίσως. Σχετικά με τις δικές μου τροπολογίες, πόνο 12, με συγχωρείτε κύριε Στρέλα, που τόσες κατέθεσα έχει να κάνει με την παρεχώρηση και για τη διαχείριση ακριβώς αυτή και τον ορισμό που έχει να κάνει όλα αυτά με την ορολογία της οδηγίας και τη σχετική σύνταξης. Αυτός ο ορισμός για την ε, συμφωνία της σύμβαση που λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτή η ανταλλαγή και με θετικά σημεία και για τις δύο πλευρές ε, για ορισμένους ε, κινδύνους ζήτησης προσφοράς αυτό θα πρέπει και τα δύο συμβαλόμενα μέρη να τα προστατεύσει σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης και εκείνο που λαμβάνει και επίσης για τα 5 εκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαν να δοθούν χωρίς ε, διαγωνισμό και επίσης ε, όλα τα στοιχεία τα τεχνικά που μπορούν να ισχύσουν όπως επίσης και τα οικονομικά και ε, αυτό το έγγραφο παραχώρησης που είναι μαζί και με την προκήρυξη. Θα ήθελα να κάνω δύο επιπλέον να δώσω ας το πούμε συμβουλές, ε, υποδείξεις ε, ότι θα πρέπει την αρχή της επικορικότητας να τη σεβόμαστε. Οι τοπικές αρχές, οι τοπικοί φορείς θα πρέπει να είναι πάντα ελεύθεροι αν ε, θα το κάνουν όλο αυτό μόνοι τους είτε θα το παραχωρήσουν το έργο σε τρίτους και σε περίπτωση αυτή η εκτέλεση σε τρίτους θα πρέπει να καθορίσουν το νομικό μέσο το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί με μία άδεια παραχώρηση, δημόσιο διαγωνισμό, οτιδήποτε και εναπλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, το είδαμε αυτό, δηλαδή ε, με μια πιστοποίηση κατάλληλη που αποτελεί τις περισσότερες φορές μια μεγάλη απλούστευση και όσον αφορά την ε, ε, ανάθεση τελικά και όλοι εποφελούνται και χρονικά και οικονομικά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν. Παρακαλώ όμως να είναι πολύ σύντομη, γιατί ήδη έχουν καθυστερήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότηση. Να εξηγήσω δύο-τρία κύρια σημεία που έθιξε ο εισηγητή και οι ομιλητέ. Να σας διαβεβαιώσω ότι η οδηγία αυτή δεν στοχεύει ούτε στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών, ούτε στον περιορισμό της ελευθερίας των δημοσίων αρχών να αποφασίσουν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να χορηγούν κάποιες δημόσιες υπηρεσίες. Το λέει μάλλον σαφέστερα, το διευκρινίζει ακόμη περισσότερο. Δεν υπονομεύει λοιπόν αυτές τις αρχές, το αντίθετο υπάρχει. Επίσης πλήρες ελευθερία στα κράτη-μέλη να καθορίζουν τις ε, κοινέ υπηρεσίες, Τη υπηρεσία γενική κοινή ωφέλεια. Είναι θέμα κράτου μέλους. Εισάγει διαφάνεια όμως, όχι διακρίσει, στι δημόσιε προμήθειε και ισότιμη μεταχείριση. Επειδή οι δημόσιε προμήθειες ε, είναι στα πλαίσια της ευρύτερη δαπάνη δημοσίου χρήματο, χρειαζόμαστε λοιπόν κανόνε, να διασφαλίσουμε λοιπόν και την ίση μεταχείριση και ότι υπάρχει νομική ασφάλεια για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αυτές οι συμβάσεις από τις δημόσιες αρχές. Τελευταίο, η οδηγία αυτή αφήνει αρκετό χώρο, άνετο χώρο, για να συμπεριληφθούν κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Δεν υπονομεύει καθόλου την ε, νομοθεσία, τη δευτερογενή νομοθεσία στον τομέα των δικαιωμάτων εργασομένων. Και βεβαίως ε, είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω επεξεργασία του κειμένου αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. 9 ε, Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε. Τελευταίο σημείο, ακρόαση. Χαιρετίζω τους προσκεκλημένους μας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Έχουμε μία ακρόαση για τις επαγγελματικές ασθένειες ε, λόγω του αμοιάντου και τις προοπτικές εξάλληψης έχουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας που είναι η βάση της πρωτοβουλίας αυτής. Θα τη συζητήσουμε ε, στις 9 Οκτωβρίου και δίνω το λόγο πρώτα απ' όλα στον εισηγητή μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο, διότι ήδη έχουμε καθυστερήσει σε σχέση με την προβλεπόμενη ώρα έναρξη τη ακρόαση. Η πρώτη έκθεση που συνέταξα για το θέμα του Αμιάντου ήταν και η πρώτη μου έκθεση γενικότερα με την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή. Πολλά χρόνια πριν. Ο Άλεξ Φόλκνερ από την Σκοτία, ε, δούλευε στα ναυπηγεία στην ε, Σκοτία και ε, προσευλήθη από την αμοιάντωση, την ασβέστωση και τελικά πεβίωσε. Δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο έκθεσης. Αυτό θέλω να καταλήξω. Αυτή η ουσία είναι θανατηφόρα και φέρνει το θάνατο 30-40 χρόνια μετά την έκθεση. Είναι παραταταμένη η περίοδος ανάπτυξης ε, της νόσου. Τώρα βεβαίως γνωρίζουμε πολλά περισσότερα για αυτήν την ε, νόσο και έχουν απαγορευτεί από τη θέση σε εμπορία και τη χρήση ε, διάφορα μιαντούχα υλικά. Επίσης θεσπίσαμε διάφορες οδηγίες για να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους που εκτίθενται στον αμίαντο και πλήττονται από αυτούς τους κινδύνους που συνεπάγεται η αφαίρεση και η ασφαλής μεταφορά του υλικού. Έχουμε ρυθμίσει αυτό το πρόβλημα, όμως εκκρεμούν και τα ζητήματα το κυριότερο των οποίων είναι ε, τώρα που ισχύει η απαγόρευση εξακολουθούμε να έχουμε εκατομμύρια τόνους ε, στα πλοία, στα τρένα, σε κτίρια, δημόσια ή και ιδιωτικά, σε σχολεία, σε νοσοκομεία. Υπάρχει υψηλότατο κίνδυνος ακόμη και σήμερα ε, μαθητές στο σχολείο να εκτεθούν ε, και οι ίνες μπορεί να οδηγήσουν σε διάφορες ε, ασθένειες όπως το μεσοθυλίωμα, η ασβέστοση και να οδηγήσουν στο θάνατο. 20 με 30 χιλιάδες περιπτώσεις διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στην στο ανώτατο ε, αριθμό κρουσμάτων ε, θα χειροτερέψει η κατάσταση τα επόμενα χρόνια. Παρά την απαγόρευση δεν υπάρχει αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου ε, των εισαγωγών των ιαμιαντόχων υλικών. Έχουμε τρία κράτη-μέλη που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τη σχετική απόκληση που επιτρέπει την περιορισμένη χρήση του ε, αμύαντου σε εξοπλισμό αιμοκάθαρσης, ε, παραδείγματος χάρη, ε, ενώ έχει απαγορευτεί γενικότερα η χρήση αυτού του υλικού στην, για όλο τον εξοπλισμό. Θα ήθελα τώρα να σας εκθέσω την θέση μου με την, ως εισηγητής. Δεν υπάρχει ε, ασφαλές επίπεδο έκθεσης ε, στον αμίαντο. Έχουμε ε, μεγάλες ποσότητες αμίαντου σε διάφορες υποδομές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πολύ διαφορετικά επίπεδα κατάρτισης που προβλέπονται στα διάφορα κράτη-μέλη για τους εργαζόμενους που έρχονται σε επαφή με τον αμίαντο, κυρίως στον τομέα των ανακαινήσεων. Οι εργαζόμενοι εκτίθενται στον αμίαντο και όσο περισσότερος χρόνος περνάει με μετά την ε, θέση σε εφαρμογή του της απαγόρευσης, ε, τόσο λιγότερο πιθανό είναι οι εργαζόμενοι να γνωρίσουν ότι πρόκειται για μια, όταν τελικά έρθουν σε επαφή με το υλικό. Τώρα ε, η ολική, η μερική αφαίρεση, ο εγκλισμός του Αμοιάντου. είναι δραστηριότητες που αναλαμβάνουν κάποιες εταιρείε ανακαίνεση, Γνωρίζουν ακριβώς πού είναι ο Αμίαντο. όμως δεν υπάρχει χαρτογράφηση του τοπίου. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς ε, πού ε, ενδέχεται οι εργαζόμενοι να εκτεθούν στον αμύαντο. Είπα ότι θα είμαι σύντομος, ήδη έχω μιλήσει υπερβολικά πολύ. Θα ήθελα ε, ε, τηλεγραφικά να αναφερθώ στους, ε, στα βασικά κεφάλαια της έκθεσής μου, δεξιότητες και κατάρτιση. Σας είπα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ισότητα ως προς την κατάρταση που προσφέρεται, αφαίρεση τώρα, καλύτερη χαρτογράφηση του, του για αποτελεσματικότερη αφαίρεση, να ασχοληθούμε με τις ευπαθέστερες ομάδες, δηλαδή υπάρχουν ενώσεις των θυμάτων που ήδη εργάζονται σε μεγάλο βαθμό για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, αλλά δεν την χάνουν υποστήριξη. Επίση, ε, δεν ξέρω αν έχετε δει τι εικόνε από ε, νέου εργαζομένου, από παιδιά ε, ε, που εργάζονται στο Μπαγκλαντές, ε, στην Ινδία, σε ναυπηγεία, επισκευάζοντας πλοία που είναι γεμάτα από αμύαντο και εκρήθενται καθημερινά. Και ε, γενικότερα στις τρίτες χώρες συμβαίνει αυτό τώρα θα προσπαθήσουμε να εξωστρακίσουμε παγκοσμίω ε, τον αμύαντο, να ενθαρρύνουμε και άλλες ε, χώρες, να δείξουμε ποια βήματα έχουμε ήδη κάνει εμείς για την απαγόρευση της χρήσης του υλικού, αλλά ξαναλέω ότι εκκρεμού ζητήματα δεν έχουν ρυθμιστεί όλα. Τέλος, μόλις μίλησα με έναν ε, Γερμανό δικηγόρο, πρωτού μπούμε στη συνεδρίαση και εκπροσωπεί εργαζόμενους που έχουν εκτεθεί στον αμύαντο και μου θύμισε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πρόκειται μόνο για τους εργαζομένους, αλλά πρόκειται και για τις οικογένειές τους ε, συχνά. Ε, εσχάτως υπήρχε μια περίπτωση ενός ε, μηχανικού που εγκαθιστούσε καλώδια σε σωλήνες που περιείχαν αμίαντο και σε μία μόνο στιγμή έκθεση της γυναίκας αυτού του ανθρώπου στον αμίαντο προσευλήθη από το την όσα θα σταματήσω να μιλάω εδώ και θα αφήσω τους εμπειρογνώμων να μας ε, αναλύσουν το ζήτημα. Σας ευχαριστώ, λέει η Προεδρεύουσα. Θα ήθελα τώρα να σας ενημερώσω ότι μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τους εμπειρογνώμονε καθώς και τις παρουσιάσεις τους φακέλους που έχουν μοιραστεί. Ας ακούσουμε τώρα α, τους εμπειρογνώμονες 10 λεπτά έκαστος. Ε, η κυρία Κρίστα Ζέτλατσεκ ε, θα πάρει πρώτα τον λόγο. Καλώ ορίσατε. Είστε η Διευθύντρια ε, ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω μια αίσθηση déjà vu γιατί η σχέση μου με τον αμίαντο Άρχισε το 1983, μόλις τελείωσα τις σπουδές ε, ιατρική, πήγα στην επιθεώρηση εργασίας και μεταξύ 83-90 στην Αυστρία πάλεψα για την απαγόρευση του αμοιάντου, έγιναν πολλές συναντήσεις, υπήρξαν ε, εμπειρογνωμοσύνες πολύ διαφορετικές και επίμαχες. Σε αυτά τα 7 χρόνια, 83-90, επιβάλαμε την απαγόρευση αυτή και το 92 το δέχτηκε και η Γερμανία και το 95 σε επίπεδο ένωσης. Όπως Στίβεν είπε ήδη, αυτό δεν σημαίνει πως έχουμε δει το τέλος αυτού του προβλήματος. Η κατάσταση είναι ασταθής στην Αυστρία γιατί κάποιες ε, εταιρείες παράγουν τσιμέντο από αμίαντο για κάλυψη των στεγών. Βεβαίως υπάρχουν πολύ σοβαρά μέτρα ε, ασφάλειας για τη χρησιμοποίηση αυτού του υλικού, αλλά το επικίνδυνο είναι ότι υπάρχει τεράστιος χρόνος λανθάνουσας ε, ύπαρξης της ασθενείας, μπορεί μέχρι 40-50 χρόνια. Και είναι και ιδιαίτερα απρόβλεπτο που μπορεί να προκύψουν αυτά τα προβλήματα, όπως είπαμε, σε εργασίες συντήρησης ή καθαρισμού. Είμαι λοιπόν ε, διευθύντρια του οργανισμού αυτού, αλλά δεν θέλω να θυμίσω μόνο αυτή την περίοδο 83-90, όταν συζητούσαμε την ε, συνολική απαγόρευση, αλλά από τη στιγμή εξόριξης μέχρι τελικής αποθήκευσης του αμοιάντου δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζει κανείς ποτέ τον αμοιάντο με ασφαλή τρόπο. Εδώ βλέπετε δύο πνεύμονες. Αριστερά ένας φυσιολογικός πνεύμονας, δεξιά ένας ε, πνεύμονας που έχει θυγεί από καρκίνο και αμιάντωση. Βεβαίως ε, ο αμύαντο έχει θαυμάσιες ιδιότητε Είναι ένα υλικό πυρητιώδε το οποίο είναι οι που υπάρχει και στο περιβάλλον, αλλά και μέσα στους, ε, αλλά και μέσα στους ε, ιστούς και μέσω εισπνοής αποθηκεύεται και το ανοσοποιητικό σύστημα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις ίνες. Δημιουργούνται λοιπόν ε, πληγές και τελικά δημιουργούν τέτοια προβλήματα στην αναπνοή που μειώνεται η πρόσληψη οξυγόνου και δεν μπορεί κανείς του καν να περπατήσει. Και επίσης μπορεί να προκύψει και καρκίνος ε, το μεσοθυλίωμα, διάφορες άλλες μορφές καρκίνου. Μπορεί επίσης να έχουμε και καρκίνο του στομάχου, του εντέρου και έχει επίπτωση και στις καρδιοαγγειακές ασθένειες. Όπως είπα και προηγουμένως, οι θαυμάσιες ιδιότητες ε, του αμοιάντου μπορεί να αντιμετωπίσει πολύ πίεση, θερμότητα, είναι πολύ καλό μονοτικό υλικό. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι στην περίοδο μεγάλης οικονομικής ε, ανάπτυξης μέχρι το 1995 σε όλους τους τομείς χρησιμοποιήθηκε. Οπότε έχουμε αυτό το άκθος του παρελθόντος σήμερα όπου χρησιμοποιήθηκε άσβεστος πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το υλικό βεβαίω σε πολλά κτίρια, σε πολλά πλοία και συνολικά στην ε, βιομηχανία Χάλιβα χρησιμοποιείται σε καταστάσεις της βιομηχανίας Χάλιβα για προστασία κατά της πυρκαγιάς και επίσης στα κεραμικά και επίσης στα ελαστικά βάζαμε παλιότερα αμίαντο είναι αυτό το παλιό άχθος. Σήμερα λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια εργασία εξυγίανσης και τις εργασίες καθαρισμού, τις εργασίες διάλυσης, τις εργασίες απόθεσης. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το πρόβλημα αυτό. Όλη αυτή η αλυσίδα, όλες αυτές οι εργασίες πρέπει να γίνονται με πολύ μεγάλη προσοχή. Βεβαίως υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν ε, οδηγίες χρήσης, αλλά ασφάλεια 100% δεν υπάρχει. Επιπλέον, πρέπει να ξέρετε ότι εισάγουμε από την Κίνα και τη Ρωσία αμίαντο όπου εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε χωρίς κανένα περιορισμό. Εισάγουμε προϊόντα που τον περιέχουν τι κάνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία μου. Το 2003 είχαμε τη δήλωση της ε, Δρέσδης, στην οποία συμμετέχουμε από το 2003 και εμείς, που προβλέπει πολλά μέτρα προστασίας όταν εργαζόμαστε με προϊόντα που περιέχουν αμίαντο. Έχουμε κάνει δύο καμπάνιες για το θέμα αυτό. Το 2004 ασχοληθήκαμε με το κατασκευαστικό τομέα όπου βεβαίως μιλήσαμε και για τον αμίαντο και το 2010 κάναμε μία καμπάνια δύο ετών όπου ασχοληθήκαμε με τις εργασίες συντήρησης και επίσης παραγάγαμε και πολλά υλικά που είναι και στο site μας όπου προσπαθούμε όπως υπόθηκε και πριν να καθιστούμε κατανοητά τα θέματα αυτά και προσπαθούμε να έχουν και εύκολα πρόσβαση. Συμμετείχαμε επίσης στην καμπάνια των ανωτέρων ε, εποπτικών αρχών για θέματα ασφαλείας και υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμβάλαμε και εδώ λοιπόν και, ανα... και ε, εκπονήσαμε υλικά όπου λοιπόν συμμετέχουν επιθεωρήσεις εργασίας από όλα τα κράτη-μέλη υπάρχουν κάποια προβλήματα να δούμε πού ακριβώς υπάρχει αμίαντος μετά από αυτή την καμπάνια είπαμε σαφώς ότι δεν μπορούν μόνοι οι επιθεωρητές εργασίας να ασχοληθούν με το θέμα αυτό. Πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι, οι συνδικάτα, εργοδότες να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό. Για παράδειγμα, ήδη αναφέρθηκε, οι νέοι εργαζόμενοι, για παράδειγμα, στο κατασκευαστικό τομέα δεν έχουν δει ποτέ αμίαντο. Μόνο και μόνο δηλαδή να τον αναγνωρίσουν. Είναι δύσκολο. και δεν ε, έχει κανείς υπόψη του ακριβώς ποια είναι αυτά τα προϊόντα που περιέχουν. Δεν είναι εύκολο να τα αναγνωρίσει τα προϊόντα που περιέχουν αμίαντο. Ορισμένε φορές δεν φαίνεται ο αμίαντο. Στις εργασίες ανακαίνησης και συντήρησης επίση πρέπει να έχουμε τις σωστές διαδικασίες. Πρέπει να γίνεται αποτίμηση του κινδύνου που δεν γίνεται πάντα ή σε πολύ μικρό βαθμό. Και τι μέτρα τα μέτρα ορισμένε φορέ δεν εφαρμόζονται με τον σωστό τρόπο, με τι σωστέ μεθόδου. Κατά την διάλυση και μετά μεταφορά και εναπόθεση του αμοιάντου έχουμε μεγάλα προβλήματα για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, διότι δεν υπάρχει σωστή κατάρτιση των εργαζομένων γι' αυτό. Και οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τέτοιου τύπου εργασίες δεν είναι οι πιο ενδεδειγμένες, δεν υπάρχει διαδικασία χορήγησης αδειών για τέτοιου τύπου εργασίες. Πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί η κατάσταση ενημέρωσης και διαφάνειας. Δεν είναι επαρκής. Στις ε, χώρες μέλη είναι σποραδική η έκθεση στον αμίαντο, αλλά είναι πολύ τακτική στον ε, τομέα το κατασκευαστικό και τα παρεμφερεί. Αλλά τα περισσότερα έχουν να κάνουν με την διάλυση, τη συντήρηση, εξυγίανση. Αλλά αυτό δεν αφορά μόνο τον τομέα των κατασκευών. Αφορά και την ανακύκλωση, τα τρένα, η ανακύκλωση τσιμέντου με αμίαντο ή τα εμπορευματοκιβώτια που περιέχονται τέτοια υλικά Υπάρχουν και διάφορα είδη ε, αμίαντου. Υπάρχει βέβαια το τσιμέντο μπασβέστη όπου είναι, που είναι πολύ συμπαγές, αλλά υπάρχουν άλλα είδη αμιάντου που είναι πολύ χαλαρά κολλημένα και πολύ εύκολα ε, αποκολλώνται από διάφορες καταστάσεις. Συστάσεις λοιπόν που προέκυψαν από αυτήν την ε, καμπάνια, αυτή την εκστρατεία. Σημαντικές λοιπόν πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τους εργαζόμενους για τους ενδεχόμενους κινδύνους, καλή και διαφανής ενημέρωση, εύκολα προσβάσιμη, εύκολα κατανοήσιμη από κάθε εργαζόμενο και τακτική ενημέρωση επιτόπου, εκεί που γίνονται οι εργασίες, κατάρτιση όχι μόνο για τους εργαζόμενους, αλλά και για τους επιθετές εργασίες, τους εργοδότες και επίσης να υπάρχουν επαρκείς ειδικευμένες δυνα... ε, ε υπηρεσίες ασφαλείας που να προσπαθούν να ε, βοηθήσουν. Και επίσης να υπάρχουν και οι σωστές διαδικασίες που να μπορούν να αναγνωρίζουν την παρουσία τέτοιων υλικών και διαφάνεια σωστή ενημέρωση για όλους τους εργαζόμενους. Συντονισμός επιτόπου, για παράδειγμα στα διάφορα εργοτάξια. Πρέπει λοιπόν να συμπεριληφθούν και εμπειρογνώμονες σε αυτήν την προσπάθεια και πρέπει να υπάρχει σαφής ευθύνη. Τέλος, η μεταφορά και εναπόθεση των αμιαντούχων υλικών πρέπει να είναι και σωστά σημασμένη. και για τις επιπτώσεις λοιπόν στο περιβάλλον. και όσοι επίσης ασχολούνται με απορρίμματα που περιέχουν αμίαντο κάνουν μια πολύ επικίνδυνη εργασία και σε αυτό το τομέα λοιπόν πρέπει να γίνεται αποτίμηση της επικίνδυνοτητας να καθαρίζονται σωστά όλα τα εργαλεία, να μην έχουν πάνω σκόνη που περιέχει αμίαντο και τακτική έλεγχη. Μία από τις επιπτώσεις που εξαγάγαμε και από αυτήν την καμπάνια των επιθεωρητών εργασίες Το είπα και στην αρχή. Δεν επαρκεί η επιθεώρηση εργασίας. Η... Για να ε- έχουμε βελτίωση των συνδικών εργασίας πρέπει να εργαστούμε όλοι από κοινού για την πρόληψη των κινδύνων. Αυτό είναι το πόρισμα και από αυτήν την εκστρατεία των ανωτάτων αρχών επιθεώρησης εργασίας. Όλοι πρέπει να συμμετάσχουν οι εργοδότες, τα συνδικάτα, οι εμπειρογνώμονες. Όλοι πρέπει να εργαστούμε προς την ίδια κατεύθυνση. Να αναφέρω πάλι καταληκτικά Υπάρχουν πολλοί λόγοι που συνηγορούν στην απαγόρευση του αμοιάντου. Δεν υπάρχει καμία ασφαλής χρήση του αμοιάντου 100%. Υπάρχουν καλές νομοθετικές ρυθμίσεις για όταν πρέπει να εργαστούμε με τέτοια υλικά. Όλες λοιπόν οι συνθήκες αυτές πρέπει να εφαρμόζονται. Αυτά είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω ερωτήσεις. Ευχαριστώ λέει πρόεδρος, ε, δόκτωρα Σελλατσέκ. Και τώρα έχω την ευχαρίστηση να δώσω το λόγο στον κύριο Τίμο Τουόμι. Είναι διευθυντής του Φιλανδικού Ινστιτούτου Υγείας της Εργασίας. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Εκπροσωπώ το Φιλανδικό Ινστιτούτο Επαγγελματική Υγεία. Είναι ένα Ινστιτούτο Εμπειρογνωμόνων που κάνει έρευνα και προσφέρει υπηρεσίε σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια. Θα ήθελα εντάχει να σας ε, πω ότι η εμπειρία που έχω για τον αμίαντο και για τις ε, σχετικές νόσους προέρχεται από τη διατριβή μου ε, ερευνούσα τους ασθενείς μεσοθυλιώματος μετά από έκθεση σε αμύαντο τη δεκαετία του 90. Στη συνέχεια ετέθηνε επικεφαλής του εργαστηρίου ε, που διεξήγαγε ανάλυση για τον αμύαντο. Ε, είναι, πολύ, είναι ιδανικό το μέρος για να συνειδητοποιήσει κανείς τι συμβαίνει με την υγιεινή για την προστασία από τον αμύαντο και τι συμβαίνει επί τόπου στις οικοδομές. Ίσως να αναφέρω ότι ε, βρίσκομαι εδώ διότι μετήχα στην ε, ομάδα εμπειρογνωμόνων που τα τελευταία δύο χρόνια επεξεργάστηκε ε, την εθνική νομοθεσία για το ζήτημα αυτό. Μπορώ λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μου και τα όσα έμαθα στην Φιλανδία αν αυτό μπορεί να συνεισφέρει στην συζήτησή σας εδώ. Ας αρχίσω παρουσιάζοντας ε, την κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράγεται, εξορίζεται ακόμη ε, ο αμύαντος σε 2 εκατομμύρια τόνους, ε, κυρίως στη Ρωσία, την Κίνα και άλλες χώρες και στον Καναδά συγκεκριμένα Πάρα πολλοί άνθρωποι εκτίθενται ακόμη και σήμερα και ένας ε, πάρα πολύ μεγάλος ε, αριθμός ε, ασθενών αποβιώνουν λόγω των σχετικών νοσημάτων κάθε χρόνο. Από την έρευνα και την τεκμηρίωση που έχουμε γνωρίζουμε ότι όλα τα είδη αμύαντου που αναφέρονται εδώ μπορούν να οδηγήσουν σε νεοπλάσματα, σε καρκίνους. υπάρχουν κάποιες διαφορές, αν δεν υπάρχει ασφαλής μορφή αμύαντου. Θυμηθείτε επίσης ε, ότι το ίμιση των θανάτων ε, ε, επαγγελματικού καρκίνου προέρχονται από τον αμύαντο και φτάνουμε στο 90% στην Φινλανδία. δύο στοιχεία μόνο. Εδώ ε, εξορίσατε ακόμη ο αμύαντος και ε, εδώ βλέπετε ένα ανοιχτό ρηχείο στη Ρωσία σε μικρή κλίμακα και μια, ένα στιγμιότυπο από την παραγωγική αλυσίδα δεξιά. Εμφανίζεται το αμύαντος ως ένα κονίαμα γκρι. Θυμηθείτε επίσης ότι τα ορυκτά, τα, τα μιαντούχα ορυκτά είναι οι νόδι. Αυτή είναι η βασική τους ε, ιδιότητα. Εδώ βλέπετε την εικόνα του μικροσκοπίου. Εμφανίζεται ο ε, συνόδες υλικό, το ορυκτό αυτό. Υπάρχουν ε, οριακές τιμές για την έκθεση στον αμίαντο. Ε, μετρά τη συγκέντρωση σε ίνες ανά εκατοστό του αέρα. Το να συγκρίνει κανείς ε, την οριακή τιμή ε, του καθαρού αέρα ή του αέρα που έχει καθαριστεί μετά από αφαίρεση αμοιάντου. Ε, περνάμε από το 4,3 στο, ε, στη 0,1 είναι ένα κυβικό εκατοστό του αέρα. Ε, που ε, υπάρχει έκθεση στο χώρο εργασίας, στον ε, περιβάλλοντα αέρα, στα εργοτάξια, σε χώρους κατεδάφισης που δεν, όπου δεν ελέγχεται η σκόνη και μεταφέρεται παντού. Ή, παραδείγματο χάρη, ένα φορτηγό που μεταφέρει απορρίμματα που περιέχουν ε, αμίαντο, μεταδίδει επίσης δια το αέρος ε, τον αμίαντο. Επίσης, ε, ο αέρας στο εσωτερικό των κτηρίων μπορούν να ε, να ε, έχουν επίσης ένα εύθρυπτα υλικά μία του. Ε, οι ίνες συγκεντρώνονται δε στους πνεύμονες των ασθενών και παραμένουν μακροχρόνια εκεί για το υπόλοιπο της ε, ζωής τους για δεκαετίες ολόκληρες έχουν τις ίνες οι ασθενείς στους πνεύμονές τους και ε, είναι χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνεται η νόσος ε, πολύ αργότερα από, την πρώτη, από τη στιγμή της πρώτης έκθεσης. Ο προλαλής σας ε, αναφέρθηκε στη, στα νοσήματα, στις, στους διάφορους καρκίνους, δεν χρειάζεται να επαναλάβω κι εγώ. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα για την έκθεση στο χώρο εργασίας ή στο εσωτερικό των κτηρίων. Η έκθεση συμβαίνει στο χώρο εργασίας, σε χώρο ελεγχόμενο, το χώρο της οικοδομής. Όταν ε, ο αμύαντος έχει παραμείνει μέσα σε συσκευές ή μέσα στα κτίρια γενικότερα, όσοι ασχολούνται με την συντήρηση των εγκαταστάσεων ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, νερού ή θέρμανσης, δυστυχώς μπορούν να εκτεθούν. Επίσης το θέμα της παράνομης εναπόθεσης και αποθήκευση αμύαντου σε χωματερές επίσης παράνομα απόβλητα μπορεί να περιέχουν αμύαντο σε εργασίες εξκαφής επίσης υπάρχει κίνδυνος έκθεσης όταν μιλάμε βεβαίως για την ατμόσφαιρα και για το, το εσωτερικό των ε, κτηρίων. Όπως σας είπα προηγουμένως, ε, υπάρχουν πολλοί που είναι εκτεθειμένοι. Στη Φιλανδία, παραδείγματο χάρη, έχουμε αφαιρέσει περίπου 50% και το 50% παραμένει. αποτυχημένος έλεγχος ε, της ε, σκόνης ε, ή το να μην λαμβάνουμε υπόψη το θέμα του αμύαντου όταν γίνεται κάποια συντήρηση, μετατροπή ή κατεδάφιση μπορεί να οδηγεί σε μεγαλύτερη έκθεση των εργαζομένων. Συνοπτικά θα έλεγα ότι είναι δυνατόν να γίνει με ασφαλή τρόπο η αφαίρεση ε, του αμοιάντου. Από τεχνικής πλευράς έχουμε επαρκείς γνώσεις, ε, καλές πρακτικές, ε, μεγάλη εμπειρία ως προς το τι πρέπει να κάνουμε. Όμως κατάρτιση, ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία είναι πράγματα που θα χρειαστούμε για να υλοποιήσουμε τον τελικό μας στόχο, την ε, ολική αφαίρεση του Αμμιάντου. Συνέλεξα διάφορες ε, προτάσεις και συστάσεις που προέκυψαν από την ομάδα εργασίας που προανέφερα όταν επεξεργαζόμασταν ε, το σχετικό φιλανδικό νομοσχέδιο και καταλήξαμε στο ότι σημείο κλειδί είναι και πάλι οι δεξιότητες οι εργολάβοι, οι εργοδηγοί ε, πρέπει να είναι σωστά ενημερωμένοι και κατηρτισμένοι για να μπορέσουν να προστατευτούν οι εργαζόμενοι. Το ίδιο ισχύει και για όλους τους εμπλεκομένους. Επίσης, ε, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σωστά κατηρτισμένοι επαγγελματίες για την αφαίρεση του αμοιάντου Επίσης θα πρέπει η κάθε μονάδα επαγγελματικής υγείας, υγείας στον χώρο εργασίας να παρακολουθεί στενά την διαδικασία, να δίνει σωστές συμβουλές, να ενημερώνει για τους κινδύνους ε, που ενέχει η έκθεση στον αμίαντο, να προτείνει τρόπους προστασίας κτλ. Επίσης ε, είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου να χαρτογραφηθεί ο αμύαντος ε, που υπάρχει ε, σε όλα τα καταλήμματα, σε όλα τα κτίρια και να ε, καταγραφούν αυτά τα στοιχεία για να αποφευθεί η έκθεση όταν, όταν γίνεται η συντήρηση, η ανακαίνιση ή η μετατροπή αυτών των κτίριων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, Mr. Tuomi, for your Ευχαριστώ κύριε Τουόμι για τη συμβολή σας. Ο επόμενος ειδήμων, ο κύριος Βέτσμαντα, είναι από... Είναι διοικητικό τέλεχο του BET e του Ινστιτούτου Υγεία και Ασφάλεια Εργασία τη Δανία. Δανική Ομοσπονδία Θεγαλιστικών Οργανώσεων Οικοδόμων. Σας ευχαριστώ. Ναι, μια και μπορώ να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα θα υποφεληθώ, ενώ είχα ετοιμάσει την ομιλία μου στα αγγλικά. Για να δούμε λοιπόν το νόημα αυτής της έκθεσης στον αμίαντο και τώρα εάν υπάρχει μια απαγόρευση, αλλά πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στο μέλλον. Εγώ διαθέτω 30 χρόνια πείρας με πολλές και διάφορες δραστηριότητες σχετικά με το θέμα του αμοιάντου. Εγώ εργάστηκα για την εγκατάσταση, για την απομόνωση, εργάστηκα σε συνεργασία με γιατρούς ε, από, την, ε, από νοσοκομείο που ασχολιόταν ειδικά με τον αμίαντο και επίση στενή συνεργασία και με ιατρούς αλλά και συνδικάτα καθώς επίσης και πανεπιστημιακούς ερευνητές. Ήταν λοιπόν ε, ένα τεράστιο όγκο δουλειά και στη Δανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με του προσανατολισμούς, τι ρυθμίσει και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Ε, και θα πρέπει να δούμε ακριβώς ε, το θέμα σχετικά με τις οικοδομές. Θα πρέπει να προσέξουμε πόσο επίγουσα η κατάσταση ε, πολλά κράτη από τη δεκαετία του 70, του δεκαετία του 80 απαγόρευαν ε, τον αμίαντο μέχρι και το 90 και 30 χρόνια πάρα πολλοί πολιτικοί, πάρα πολλοί τεχνικοί συνεργάστηκαν για την απαγόρευση του αμιάντου, αλλά χρειάστηκαν, απαιτήθηκαν 30 χρόνια. Ας μην ξεχνάμε και το κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Υπάρχουν όμως και μερικές εξαιρέσεις μια οδηγία η οποία ε, ρυθμίζει τα πράγματα για μια σίγουρη εργασία. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο μίαντος ε, είναι θανατηφόρα ουσία και σε πολλά τρένα, σε πολλά πλοία υπάρχει ακόμα και σε κτίρια και σε δημόσια και σε ιδιωτικά. οι αριθμοί για τον αμίαντο δεν είναι πάντα αξιόπιστοι. Πολλές φορές το περιεχόμενο σε αμίαντο είναι υψηλότερο και υπάρχει και ο παράγοντας χρόνος. Ο χρόνος είναι εις βάρος μας. Θα πρέπει να μπορούμε να αφαιρούμε όσο γίνεται πιο σίγουρα τον αμίαντο εκείνοι που εγκατέστησαν υλικά με αμίαντο και γνωρίζουν πώς να τον αφαιρέσουν ε, συνταξιδοντούνται τώρα. Άρα λοιπόν η νέα γενιά στον τομέα της οικοδομής που θα πρέπει να ασχοληθεί με την αφαίρεση του αμιάντου δεν διαθέτει τόσο πολλές γνώσεις γιατί στα νέα κτίρια δεν χρησιμοποιείται ο αμίαντος και διαθέτουν ελάχιστη πείρα επαναλαμβάνω γιατί ο αμίαντος κάποτε κάποτε κάποτε ήταν σε χρήση. Αναφερόμαστε ιδιαίτερα στην ανάγκη μιας ε, συντονισμένης στρατηγικής, ε, συνολικής σφαιρικής στρατηγικής για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα του αμίαντου. Χρειάζεται να διευρύνουμε ακόμα περισσότερο τις υποχρεώσεις για πολλές ομάδες εργαζομένων ε, που δεν καλύπτονται από την οδηγία, κυρίως στην ε, σηκοδομές και θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια εκτίμηση να δούμε ποιοι κανόνες θα πρέπει να ισχύουν για όλες τις ομάδες υψηλού κινδύνου και θα πρέπει να αναγνωριστούν οι επαγγελματικές ασθένειες που οφείλονται στον αμίαντο και ότι είναι υψηλού επαγγελματικού κινδύνου. Επίσης Υπάρχουν ακόμη τρεις χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν αμίαντο για χλωριούχα παράγωγα και σε άλλες χώρες που ισχύουν εξαιρέσεις και κυρίως τα πλοία που πουλούνται στην Ινδία και σε άλλες χώρες χρησιμοποιούν ακόμα αμίαντο παρόλη την ευρωπαϊκή απαγόρευση. Και κάτι ακόμα θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι ελπίζουμε ότι στο άμεσο μέλλον ο αμίαντος ε, θα παίξει ιδιαίτερο ρόλο με την απαγόρευσή του στον χώρο εργασίας ε, στα πλαίσια της ε, εισήγησής της για το 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συμπεριλάβει και τον αμίαντο. Χρειάζονται πολιτικές ενέργειες ε, με συγκεκριμένες προθεσμίες ε, για πότε θα μπορούσε επιτέλους ο κόσμος να ελευθερωθεί από την παρουσία αμίαντου. Χρειάζεται να κάνουμε και μία εκτίμηση. Πώς θα εφαρμοστεί η όλη νομολογία κυρίως ε, στον τομέα των οικοδομών. Και στο παρελθόν δείχτηκε αρκετά αυστηρό το κοινοβούλιο απέναντι σε χρήσεις αμίαντου και προσέχοντας τη στρατηγική περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρότρινε την Ευρωπαϊκή Τροπή να οργανώσει μια κρόαση για το πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του αμοιάντου και επίσης η Επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη σε προγράμματα δράσης σε εθνικό επίπεδο για τον αμοιάντο. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να ισχύσει, να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στα πλαίσια της νέας στρατηγικής που σε ένα-δύο μήνες θα παρουσιάσει στην κοινή γνώμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται να συμπεριληφθεί και αυτό περί αμιάντου και να υπάρξουν ε, αποτελεσματικά σχέδια, μια πραγματική εκπαίδευση, προετοιμασία και να ξέρει κανείς που υπάρχει ακόμα αμιάντος κυρίως σε παλιές βιομηχανικές μονάδες ή κατοικίες ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί με ασφάλεια. και όχι μόνο σε περιπτώσεις που ένας πολίτης ε, αποφασίζει να ε, ανακατασκευάσει το διαμέρισμά του. Χρειάζονται ιδιαίτερα βήματα και με πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου επίσης και θα πρέπει να προσέξουμε το όλο θέμα της εκτίμησης της καταστάσεως για την παρουσία αμοιάντου. Χρειάζονται και πολιτικά και τεχνικά σχέδια, αλλά χρειάζεται και η γνώση, να ξέρουμε πού ακριβώς συνεχίζει να υπάρχει αμίαντος. Υπάρχει σε πάρα πολλά κτίρια με προγράμματα δράσης και το θέμα του αμιαντού να ενταχθεί σε άλλες ε, κοινέ πολιτικές όπως την ενεργειακή ας πούμε πολιτική, την αποτελεσματικότητα την ενεργειακή των κατοικιών μας. όποιος ασχολείται με αυτά για την αριακή επάρκεια για τα κτίρια μας θα πρέπει οι εργαζόμενοι εκεί να εκπαιδεύονται κατάλληλα για να προστατεύονται από τον αμίαντο και οι ιδιοκτήτες κατοικιών ή διαμερισμάτων επίσης θα μπορούσαν να παίξουν ένα θετικό ρόλο, σημαντικό ρόλο. Υπάρχουν μητρώα σχετικά με τον αμίαντο αλλά και πάρα πολλές περιπτώσεις ε, που αγνοούν την ύπαρξη αμοιάντου οι ιδιοκτήτες. Και στα πλαίσια αυτής της ευρύτερης εκπαίδευσης ε, για την προστασία από τον απίαντο, βασικό είναι να προετοιμαστούν κατάλληλα, να εκπαιδευτούν κατάλληλα και οι αυτοαποσχολούμενοι και οι εργαζόμενοι σε εταιρείε, όλοι εκείνοι που εργάζονται στον κλάδο. Χρειάζεται συγκεκριμένο σχέδιο και μάλιστα με προθεσμίες για την αφαίρεση του συνόλου του αμίαντου. Θα πρέπει να καθορίσουμε μια ημερομηνία της πλήρους απαλλαγής από το υλικό αυτό σε όλη την Ευρώπη τα αποτελέσματα της έκθεσης των αμίαντο θα τα διαπιστώσουμε μόνο μετά από 20-30 έτη. Γι' αυτό λοιπόν από τώρα θα πρέπει να εργαστούμε για να αποφύγουμε και τον επόμενο ακόμα αιώνα να εμφανίζονται ασθένειες, συνέπειες της παρουσίας αμοιαντού και επίσης η βοήθεια στα θύματα του αμίαντο. Μιλήσαμε για τοξικά απόβλητα με αμίαντο. Χρειάζεται μια πραγματική σκληρή δουλειά για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό στην Ήπειρό μας. Τα συμπεράσματά μου λοιπόν είναι ότι χρειαζόμαστε μια εξέταση του θέματος για κατάλληλες ρυθμίσεις που να είμαστε αρκετά πρωτοπόροι με σημαντική πρόοδο στον τομέα αυτό. Μια κατάρτιση και μια ενημέρωση επαρκής αποτελεσματική, όπως επίσης και έλεγχη αποτελεσματική και η ίδια κοινή γνώμη να γνωρίζει πως έχει κατάσταση. Έχει σημασία για όλους στην Ευρώπη και επαναλαμβάνω μια προθεσμία, μια ημερομηνία που θα πρέπει πια η Ευρώπη να είναι ελεύθερη από την παρουσία αμοιάντου. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Παρουσίασή σας. Τώρα η κυρία Λόρι Κάτσεν Άλλεν, χαίρομαι για την παρουσία σας, είναι συντονίστρια του, της γραμματείας του Διεθνούς Κινήματος για την απαγόρευση του αμοιάντου στον Ηνωμένο Βασίλειο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας απασχόληση και κοινωνικών υποθέσεων που με κάλεσε να συμμετάσχω σε αυτή τη σημαντική συνάντηση. Είναι η δεύτερη ακρόαση για τον αμίαντο που έχω παρευρεθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Η πρώτη έγινε στη Βραζιλία το θέμα ήταν μια υπόθεση ενωπίων του Ανωτάτου Συμβουλίου για τη συνταγματικότητα του νόμου που επιτρέπει τη χρήση αμοιάντου στην ε, Βραζιλία. Το Σύνταγμα ε, της Βραζιλίας λέει ότι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να ζουν μια υγιή ζωή. Πώς μπορεί λοιπόν ένα αποδειγμένα τοξικό προϊόν να επιτρέπεται. Αυτό το θέμα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, τονίζει το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην ακαιρεότητα των ατόμων και το δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δηλώνει σαφώ ότι όλοι έχουν δικαίωμα στη ζωή και αυτό θα πρέπει να προστατεύεται από τον νόμο. Και παρόλα αυτά, χιλιάδε άτομα πεθαίνουν από ε, ασθένειε λόγω του αμύαντου δεν μπορούμε να ξέρουμε πού ακριβώς είναι γιατί δεν έχουμε στοιχεία από πολλές χώρες μέλη. Αυτό καθεαυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει λοιπόν κενό ενημέρωση. Οπότε έχουμε εκτιμήσεις από επιδημιολόγους που μέσω των στοιχείων για την θνησιμότητα μέσω θηλιώματος ως βάση και προσθέτοντας και τα στοιχεία για θνησιμότητα από άλλες ε, ασθένειες που σχετίζονται με τον αμίαντο. Δεν είναι παράλογο να ισχυριστούμε ότι στη Δυτική Ευρώπη μόνο πάνω από μισό εκατομμύριο άτομα θα πεθάνουν από ασθένειες που συνδέονται με τον άζωστο από το 1995 μέχρι το 2029. Επαναλαμβάνω, μισό εκατομμύριο άτομα. Αυτό θα ήταν σαν να εξλοθρευόταν ο πληθυσμός του Σέφιλ, της Γρενόμπλε, της Νιρεμβέργης και της Μπολόνια. Σήμερα μου ζητήθηκε σε 10 λεπτά να επικεντρωθώ σε κάποια ε, θέματα. Είναι δύσκολο καθήκον, αλλά επειδή έχω κάνει πολλές εκστρατείες για την απαγόρευση του αμοιάντου, έχω αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις. Πρέπει να καταλάβουμε την ανθρώπινη διάσταση της τραγωδίας του αμοιάντου στην Ευρώπη και να αντιμετωπίσουμε τις ασθένειες που σχετίζονται με τον αμίαντο. Ας αρχίσουμε λοιπόν με την ανθρώπινη διάσταση. Έχει απογρευθεί από το 2005 ο αμύαντος στην Ευρώπη. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε ασφαλείς. Αναμφίβολα όλοι μας έχουμε αμίαντο στους πνευμονές μας. Αν είμαστε τυχεροί δεν θα αναπτύξουμε ασθένεια που να σχετίζεται με τον αμίαντο. Αλλά για τους άτυχους ε, οι προοπτικές είναι σκοτεινές στις διάφορες χώρες μέλη. Αυτά που θα πρέπει να λαμβάνουν και αυτά που λαμβάνουν οι ασθενούντες από τέτοιες ασθένειες ποικίλουν πολύ. Πολλοί που έχουν ε, εκτεθεί στο σπίτι τους, στον τόπο εργασία τους ή στον αμίαντο δεν βοηθώνται επαρκώς. Το ίδιο ισχύει και για τους αυταποσχολούμενους και πολλούς που έχουν ήδη αμίαντο ε, ε, ασθένειε των πνευμόνων που σχετίζονται με τον αμίαντο. Πρέπει όλα τα θύματα αυτά να λαμβάνουν την αναγκαία στήριξη. Αλλά δεν τη λαμβάνουν. Και αυτό είναι κατά των αρχών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύσταση. Πρέπει να υπάρξει νομοθεσία που να καθιστά υποχρεωτική την τήρηση των ε, προδιαγραφών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον αμίαντο και των ασθενείων που προκαλούνται από τον αμίαντο ανεξάρτητα από τον τρόπο έκθεση των αμίαντο. Λείπουν κάποια στοιχεία στο πλαίσιο αντιμετώπισης του αμοιάντου. Μεταξύ των θυμάτων υπάρχει τεράστια έλλειψη ενημέρωσης των νομοθετημάτων και των ε, ε, συστάσεων για αντιμετώπιση του αμιάντου. Η Επιτροπή σας θα πρέπει να εγκαθιδρύσει μια υποεπιτροπή για τον αμοιάντο για να βοηθήσει την επικοινωνία μεταξύ των θυμάτων και των εκπροσώπων του στι Βρυξέλλε. Αυτή η υποεπιτροπή θα μπορούσε να επιτηρήσει τη δημιουργία ενό σώματο για να συντονίσει ένα σχέδιο δράση για τον αμύαντο στην Ευρώπη. Τμήμα τη διαδικασία αυτή θα μπορούσε να είναι ένα κέντρο για την έρευνα για τι ασθένειε που σχετίζουν τον αμύαντο. Ο ρόλο των ομάδων ε, ασθενών. Υπάρχουν πάνω από 55 ομάδε για τη στήριξη των ασθενών η γνώση αυτών των ομάδων αποτελεί μια πηγή που πρέπει να αξιοποιηθεί για όλους όσους θα πρέπει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που έχουμε έναντι των ασθενών. Πρέπει να αναγνωρίσουμε το ρόλο των, ομάδων ασθενών αυτών, να χρηματοδοτήσουμε τη δουλειά τους και να τους περιλάβουμε σε όλες τις συζητήσεις για τη μελλοντική μας πολιτική για τον αμύαντο πώς θα εξαλείψουμε τις ε, ασθένειες αυτές. Ο μόνος τρόπος είναι όλη η μας υποδομή να ε, ε, γίνει χωρίς αμύαντο. Μέχρι να το επιτύχουμε αυτό πρέπει να ληφθούν προοπτικά μέτρα για να σταματήσει η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες. Πρέπει να είναι γνωστή η ύπαρξη και ο, ακριβή ο, ακριβής τόπος όπου είναι ο αμίαντος, να υπάρχει χαρτογράφηση το που είναι ο αμίαντος και, ο, και που έχουν απορριφθεί απορρίμματα που περιέχουν αμίαντο. Οι εργαζόμενοι στον τομέα αυτό πρέπει να λάβουν υποχρεωτική κατάρτιση. Όμως ο κλάδος που ασχολείται με αυτά είναι σε χαμηλό επίπεδο και δεν έχει επαρκή επαγγελματισμό πρέπει να υπάρχει επαρκής κατάρτιση με πτυχία. Να ανεβάσουμε το επίπεδο γνώσης, να βελτιώσουμε τις μεθόδους και να προστατεύσουμε την επαγγελματική και δημόσια υγεία. Οι κυβερνήσεις πρέπει να κάνουν ε, συστηματική συλλογή στοιχείων για τις επαγγελματικές ασθένειες που σχετίζονται με τον αμύαντο, να βελτιωθεί η πρόληψη. Είναι επίσης ουσιώδες να γίνουν ε, καμπάνιες για να αυξηθεί η ε, ευαισθητοποίηση με βάση την πείρα του Ηνωμένου Βασιλείου, μια εκστρατεία που καταδεικνύει τον κίνδυνο από αμύαντο στα σχολεία θα μπορούσε να αποτελέσει μοντέλο. Δυστυχώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα περισσότερα σχολεία μα περιέχουν αμύαντο. Όλα τα είδη αμυάντου έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την οικοδόμησή του και εκτιμούμε ότι πάνω από 80% των κτηρίων που χρησιμοποιούν τα παιδιά μα κάθε μέρα περιέχουν αμοιάντο. Σύσταση λοιπόν. Η Υποεπιτροπή για τον Αμίαντο που θα εγκαθιδρύσετε θα πρέπει να έχει στόχο μια συνεκτική στρατηγική για την εξάλληψη των ασθενειών αυτών. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια προθεσμία το 2023 για να εξηγιανθεί πλήρως από τον αμίαντο η Ένωση. Να τα πρόσωπα μερικών ασθενών από αμίαντο που έχουν πεθάνει από μεσοθυλίωμα στον Ρωμανό Βασίλειο είναι το μεσοθυλίωμα, ένας καρκίνος που σχετίζεται με τον αμίαντο. Είναι μια ταχεία εξέλισης, ε, πολύ επώδυνη και θανάσιμη ασθένεια. Σκοτώνει ανελαίητα. Οι ασθενείς, τα θύματα του αμοιάντου, δεν έκαναν τίποτα κακό. Όσοι όμως επιτρέπουν τέτοιες επικίνδυνες συγκίνδυνε εργασία, οπωσδήποτε δεν είναι καθόλου ανεύθυνοι. Πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη για τα θύματα και πρόληψη μελλοντικών ασθενειών. Χρειάζεται ένα συντονισμένο πρόγραμμα και επαρκή πολιτική βούληση για την εφαρμογή του. Πρέπει να βελτιώσουμε την απόδοσή μα. Και είμαστε εδώ για να ζητήσουμε τη βοήθειά σα για να εξαλείψουμε αυτό το, την τρομερή μάστιγα, ούτω ώστε οι μελλοντικέ γενιέ να μην υποφέρουν όπω οι προηγούμενε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την συμβολή σας. Θα πρότεινα τώρα οι συνάδελφοι να έχουν δυνατότητα να θέσουν ερωτήσει, Παρακαλώ τους συναδέλφους ε, να περιοριστούν στα δύο λεπτά για να υπάρχει χρόνος μετά, για να γίνει ε, ένα κλείσιμο πέντε λεπτών από κάθε ε, έναν από τους ειδήμονές μας για να απαντήσουν και στις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ. Αγαπητέ συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να, πρέπει να πούμε στους επισκέπτες μας ότι είναι φυσιολογικό να μην είναι μεγάλη προσέλευση προς το τέλος της συνεδρίασης. Ε, πάντως ε, οι μαρτυρίες τους ε, θα διαβιβαστούν σε όλα τα μέλη της Επιτροπής και σίγουρα θα συμπεριλάβω τα στοιχεία που μας έδωσαν στην έκθεση που συντάσσω για την Επιτροπή. Οφείλω να ομολογήσω ότι συμφωνώ ως επιτοπλίστων με αυτά που μας είπαν οι εμπειρογνώμονες και τα περισσότερα ζητήματα ούτω ή άλλω αναφέρονται ήδη στην ενδιάμεση έκθεση που έχω συντάξει. όμω ε, θα ε, τροποποιήσω το σχέδιο και θα κάνω πιο αυστηρέ ε, τι προτάσει που κάνω δεδομένων αυτών των στοιχείων. 80% των σχολείων έχουν αμύαντο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μα είναι αποκαλυπτικά αυτά τα στοιχεία και σίγουρα δεν συμβαίνει αυτό μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, διότι πρόκειται για οικοδομικά υλικά που χρησιμοποιούνται σε όλη την επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να είναι και χειρότερη σε κάποια μέρη. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η καλύτερη προσέγγιση αυτή είναι και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η διάσταση. Θα το συμπεριλάβω στην γνωμοδότησή μου. Είναι ευπρόσδεκτε οι συγκεκριμένε προτάσει που κάνετε ή θα κάνετε. Θα τι ενσωματώσω στην έκθεσή μου. Ε, θα, δεν ξέρω κατά πόσο θα δεχτούν οι υπόλοιπε πολιτικέ ομάδε την πρόταση περί συστάσεω τη υποεπιτροπή, αλλά πάντω θα προωθήσουμε το θέμα εδώ, στη δική μα επιτροπή. Τέλο, πρέπει να λάβουμε υπόψη το θέμα τη χαρτογράφηση και τη ασφαλού αφαίρεση ε, του αμοιάντου στο πλαίσιο άλλων πολιτικών της Ένωσης. Ήδη έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις για την ενεργειακή αποδοτικότητα και αυτό ε, συμπεριλαμβάνει ανακαίνιση όλων ε, των κτηρίων ουσιαστικά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσαρμογή τους ε, στα νέα πρότυπα. Οπότε οπωσδήποτε μπορούμε να συνδυάσουμε το αίτημα περί χαρτογράφησης και διαδικασίας αφαιρέσης του αμύαντου. Είναι μεγάλη πρόκληση το να θέσει κανείς καταληκτική ημερομηνία για να είναι ελεύθερη αμύαντου η Ευρωπαϊκή Ένωση Μόνο ένα κράτος μέλος, η Πολωνία, έχει καταρτήσει σχέδιο δράσης και προθεσμία για να ε, επιτύχει ε, μέχρι το 2022 ολική αφαίρεση του αμύαντου. Πιστεύω ότι ε, αυτό θα έπρεπε να λειτουργήσει ως υπόδειγμα για να θέσουμε μια, ένα χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη αυτού του στόχου σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο Άντιμ και η Κρίστα σωστά έθεσαν το ζήτημα της παγκόσμιας ε, απαγόρευσης ε, του Αμιάντου. Είναι η ηθική επιταγή εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εργαστούμε προς την παγκόσμια απαγόρευση. 20 εκατομμύρια των παράγονται ακόμη στην Κίνα, τον Καναδά και τη Ρωσία, όπως ανέφεραν οι εμπειρογνώμονες. Ε, είναι ένα ζωφερό και δυσίωνο μέλλον για τις αναπτυσσόμενες χώρες, η εισαγωγή του αμοιάντου σε αυτές τις χώρες, γιατί εξακολουθεί να είναι το θαυματουργό υλικό για όπως και εμείς νομίζαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση προ δεκαετιών ε, και είναι ανήθικο, άκρος ανήθικο από πλευρά των δυτικών χωρών, διότι όσες δυτικές χώρες συνεχίζουν ε, αυτό το ε, επέσχυντο εμπόριο θα πρέπει να κατονομαστούν. Τονίζω λοιπόν την ανάγκη χαρτογράφησης να περάσει το μήνυμα ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε το, όλο το θέμα της αδειοδότης και της κατάρτισης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που εμπλέκονται στη διαδικασία αφαίρεσης και απομάκρυνσης ε, του αμοιάτου. Χρειάζεται μια συντονισμένη στρατηγική. Ακούσαμε και μια ολιστική προσέγγιση έχω ε, ε, σχετικές αναφορές στο σχέδιό μου, αλλά θα πρέπει να επαναδρομολογήσω όλα τα επιμέρους στοιχεία για να οικοδομήσω μια ε, ολιστική προσέγγιση για την αφαίρεση και απομάκρυνση του αμοιάτου, αλλά και όλα τα συναφή ζητήματα για την κατάρτιση, την ενημέρωση και την υποστήριξη προ τι ε, ενώσει που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Σα ευχαριστώ και απευθύνω και πάλι θερμή έκκληση να μα ε, συγχωρέσετε για την πτωχή προσέλευση αλλά θα διαβιβάσουμε τη μαρτυρία σα σε όλα τα μέλη τη επιτροπή. <clears throat> Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Σύντομα, σύντομα, για να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες, ε, οι οποίοι μας πρόσφεραν αυτό το πολύ ωραίο μάθημα προσπάθειας ε, ανθρώπινης για να ξεφύγουμε από αυτή την τραγωδία του αμίαντου. Να σας πω ότι με την παρουσία εδώ, επειδή δεν υπάρχουν και τόσα μέλη, αλλά παρόλα αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι. Κυρία Λάουρη, θα θυμάται ότι ήδη ε, είχαμε υποσχεθεί πολλά πράγματα και τώρα έχουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας. Εγώ από τους σοσιαλιστές ε, θα σας πω ότι όλοι οι συνάδελφοι συμφώνησαν και όλες οι ομάδες ε, κατάλαβαν τη σημασία. Είναι κάτι που προχωράει, προχωράει στην εργασία. Δεν είναι λοιπόν ανώφελη. Και εγώ θα σας πω να πω και αυτό που είπες, αυτά που είπε ο Στίβεν, ε, είναι ντροπή που τώρα, παρόλο που είμαστε σίγουροι πια επιστημονικά, επιστημονική κοινότητα, παρά αυτά, ε, ε, υπάρχει ακόμα και ακτινοβολή δυστυχώς αυτή η ουσία και για τον Καναδά. Αύριο έχουμε με την αντιπροσωπεία με τον Καναδά μια συνάντηση και θα τα μεταβάσω αυτά και με τον κύριο Χιούς ε, θα πρέπει να δούμε αυτές οι αντιπροσωπείες και κυρίως με την Κίνα, με τον Καναδά, με τη Ρωσία που συνεχίζουν την παραγωγή και μας ανησυχούν εδώ ε, με τις αντιπροσωπείες αυτές και θα δούμε, θα τα πούμε αυτά σε αυτές τις συναντήσεις μαζί τους και με πρωτοβουλίες τους συναδέλφους από εκεί να ξέρουν ότι εδώ έχουμε λάβει την υποχρέωση και θέλουμε να γίνει παγκόσμιο το μήνυμα επαναλάβω ότι σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, η προσπάθεια που εσείς καταβάνατε είναι πραγματικά ωφέλιμη. Θα αποφέρει καρπούς και μπορείτε να υπολογίζετε με εμά τους σοσιαλιστές εδώ στο Κοινοβούλιο για να συνεχίσουμε ε, τον μάχη μας, τον αγώνα μας για την δικαιοσύνη και την έλλειψη παρόμοιων ασθενειών. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ε, εμπειρογνώμονες. Δεν είμαι δήμον για τον αμίαντο. Για μένα λοιπόν ήταν πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα εισαγωγή για το θέμα αυτό. <clears throat> Συμφωνώ με τους ε, προηγούμενους. Είναι σημαντικό και επίγον το θέμα αυτό. Μία ερώτηση. Ξέρω ότι πάντα όταν ε, συντηρούμε κτίρια προσπαθούμε να μειώσουμε ε, τον αμύαντο που περιέχουν αλλά είπατε ότι το 80% των σχολικών κτηρίων περιέχουν ε, αυτό το υλικό και πολλά άλλα κτίρια. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν καταλαβαίνω ε, γιατί πρέπει να περιμένουμε τόσα χρόνια για να απαλείψουμε αυτό το υλικό. Οπότε θα ήθελα ήδη να απευθώ στα κράτη-μέλη για να ρωτήσω τι επιδοτήσει θα μπορούσαν να δώσουν στις τοπικές αρχές για να βοηθήσουν ε, την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Υπάρχουν ε, στοιχεία από τι διάφορες χώρες. Τι κόστος θα είχε για τα κράτη-μέλη εάν θα επεδίωκαν να αφαιρέσουν τον αμίαντο πλήρω από όλα τους τα κτίρια. Οπότε επανέρχομαι προς τους εμπειρογνώμονέ μας. Παρακαλώ πέντε λεπτά για να απαντήσει στις ερωτήσει μα. Σα ευχαριστώ. Δίνω πρώτα απ' όλα το λόγο στην ε, δόκτωρα Σέντλατσεκ. Ευχαριστώ πολύ. Στον οργανισμό μου και σε συνεργασία με άλλους φορείς πάντα έχουμε αυτό το ερώτημα Τι κόστος θα είχε η εξυγίανση των κτηρίων. Τι κόστος θα είχε για τους δημοτικούς φορείς. Δεν έχουμε ασχοληθεί λεπτομερώς με το θέμα αυτό. Όταν κατεδαφίστηκε το μέγαρο της ε, Δημοκρατίας στο Βερολίνο, ήμουν παρούσα και είδα τι τεράστιο κόστος είχε η κατεδάφιση και η εξυγίανση του κτηρίου. Δεν μπορώ να σας απαντήσω λοιπόν συγκεκριμένα για το κόστος. Αλλά είναι τεράστιο το κόστος για να έχουμε σωστές συνθήκες εργασίας, προστασία της υγείας. Ξέρουμε τι μέτρα χρειάζονται. Είναι τεράστιο το κόστος. Πρέπει λοιπόν ε, να ζούμε με αυτή την κατάσταση. Κάθε φορά που γίνεται κάποια συντήρηση, κατεδάφιση, προσπαθούμε να, αφαιρέσουμε τον αμίαντο Κάτι το οποίο έχει τεράστιο κόστος. Καταληκτικά. Ένα σχόλιο. Καθήκοντα ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια. Υποστηρίζουμε βεβαίως αυτές τις δραστηριότητες. Για μας ο αμίαντος είναι μια ιστορία χωρίς τέλος και τα υλικά που τον αντικαθιστούν που πρέπει να εξετάσουμε. Και βεβαίως η καρκίνη που προκαλεί προσπαθούμε στις εκστρατείες μας να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό, να αποστείλουμε ενημέρωση εργαζόμενοι μαζί με τα κράτη-μέλη, να ενημερώσουμε τις επιχειρήσεις και τους άλλους ε, απασχολούμενους στον κλάδο αυτό. Θα συνεχίσουμε αυτή μας την εργασία και σε αυτή την νέα εκστρατεία συνεργασία για αποφυγή των κινδύνων. Είναι πολύ σημαντικό η διοίκηση των επιχειρήσεων, γενικά οι εργοδότες, μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με τους ε, απασχολούμε στον τομέα αυτό να βοηθήσουν μαζί με τους επιθεωρητές εργασίες αλλά βεβαίως και ο οργανισμός αυτός κάνει αυτή την εργασία στον τομέα μας προσπαθούμε να αναπτύξουμε συγκεκριμένες μεθόδους σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη για παράδειγμα Ένα από τα εμβληματικά μας προγράμματα είναι η ηλεκτρονική αποτίμηση κινδύνων. Είναι ένα ηλεκτρονικό λοιπόν πρόγραμμα που μπορεί να βοηθήσει μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να εκτιμήσει τον κίνδυνο με πολύ απλό, μη γραφειοκρατικό, άμεσο τρόπο στο ίντερνετ. Μπορεί να το κατεβάσει κανείς αυτό το πρόγραμμα, να το χρησιμοποιήσει και βλέπουμε λοιπόν ότι στον τομέα των κατασκευών και των παρεφερών επαγγελμάτων, όπου έχουμε πολλές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ένα τέτοιο εργαλείο θα μπορούσε να βοηθήσει όλους τους εργαζόμενους με επικίνδυνες ουσίες. Θα συνεχίσουμε λοιπόν φυσικά να απασχολούμεθα με το θέμα. Έχουμε λοιπόν τα διάφορα μέσα, εκστρατείε, παροχή πληροφόρησης και ελπίζουμε να συμβάλλουμε ούτως ώστε να υπάρξει μια απαγόρευση. Αλλά το ερώτημα είναι πότε ακριβώς θα επέλθει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Λίκη Πρόεδρος. Ο κύριος Τούμι. Ευχαριστώ ε, ε, εντάχει. Ο αμύαντος πρέπει να αφαιρεθεί και θα αφαιρεθεί, αλλά το θέμα είναι η χρονική, το, η χρονική κλίμακα. Αν ε, αποσκοπούμε στην ολική αφαίρεση σε 20-30 χρόνια, αυτό ε, θα δώσει μια νέα κατεύθυνση και στην κατασκευαστική, στον κατασκευαστικό κλάδο. Δηλαδή, ένα κομμάτι της δραστηριότητάς θα μπορούσε να εστιαστεί γύρω από την αφαίρεση του αμοιάντου ε, και ένας εκπρόσωπος του κλάδου στην Φινλανδία ανέφερε ότι είναι πολύ καλή δραστηριότητα, αλλά έχει αρνητική δημόσια εικόνα και άρα δεν αναπτύσσεται αυτό το κομμάτι του κλάδου, ε, παραμένει σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ε, και το αρνητικό στοιχείο προέρχεται από την μη σταθερότητα της δραστηριότητας μικρών ε, τέτοιων εταιριών. Αν αφαιρεθεί ο αμύαντος λοιπόν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ή αν δεν αφαιρεθεί είναι τα δύο σενάρια και πρέπει να τα συγκρίνουμε από οικονομική σκοπιά. Thank you, Mr. Wittmann. Σας ευχαριστούμε, κύριε κύριος Βέτμαν. Ε, Ευχαριστώ είναι αυτό το καθήκον που αναλαμβάνουμε, δηλαδή να αφαιρέσουμε πλήρως τον αμίαντο και δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιο θα είναι το κόστος. Αυτή τη στιγμή αναπτύσσουμε ένα σχέδιο για την απογραφή τι, πού είναι το πρόβλημα όμως, είναι 20% των ε, κατοικιών ή το 80% των ε, κατοικιών, δεν ξέρω, ίσως όπως το Ηνωμένο Βασίλειο που λένε ότι είναι 80% των σχολείων. Θα πρέπει να μελετήσουμε ένα πρόγραμμα δράσης, ένα σχέδιο δράσης να δούμε το πολωνικό σχέδιο που θα κοστίσει περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2032 να αφαιρεθεί και το τελευταίο ίχνος αμίαντου. Να σας διαβεβαιώσω όμως ότι για μας είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα σε εισαγωγικά χάρτη του αμίαντου σε κάθε χώρο, σε κάθε χώρα πόσος αμίαντος παραμένει πρέπει να αφαιρέσουμε τον πιο επικίνδυνο αμίαντο. Από εκεί να ξεκινήσουμε με τους μεγαλύτερους κινδύνους λοιπόν. Εκεί που χρησιμοποιείται και είναι σε πορώδη υλικά. Ε, όχι πλήρως μεγμένο με άλλα υλικά. Και μετά να δούμε και προθεσμίες εντάξει που να ισχύσουν για μεταγενέστερη περίοδο για άλλες μορφές ε, ε, μίαντού. Πάντως ε, με αυτή την τράπεζα στοιχείων, με αυτές τις προθεσμίες ταυτόχρονα επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά θα πρέπει να έχουμε στα χέρια μας ένα χάρτη που βρίσκεται ο αμίαντος ώστε να μην έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις ε, κατά τη διάρκεια των εργασιών. Για το κόστος. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε στα πλαίσια της κρίσης της οικοδομής, η οποία έπληξε τα τελευταία 4-5 χρόνια και τη δική μου τη χώρα. Και γι' αυτό άλλαξε ιδιαίτερα η τάση όσον αφορά τις νέες οικοδομές αλλά και όσον αφορά τις ανακαινήσεις, εξυγιάνσεις ε, και λοιπά παλιότερων κτηρίων. Και εδώ υπάρχει και μία δυνατότητα ταυτόχρονα με την εξυγίαση αυτή να στα παλιότερα τα κτίρια να αφαιρούμε τον αμίαντο. Αυτά λοιπόν. Αυτό πρέπει να γίνει στο άμεσο μέλλον και χρειάζεται τρομερή προσπάθεια από πολλά κράτη-μέλη για την ε, ενεργειακή αποτελεσματικότητα, για την προστασία, για μια μόνωση όσον αφορά την τομέα της ενέργειας και η μόνωση παίζει πουδαίο ρόλο στην ενεργειακή κατανάλωση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να τα προσπαθήσουμε όλα αυτά γιατί με ένα σπάρο δύο τριγώνια θα πρέπει να κυνηγήσουμε την επάρκεια, την αποτελεσματικότητα, την ενεργειακή και τον, τον αμυαντό. Η κυρία Άλεν, να σε ενημερώσω. Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξαν εξελίξεις στην Κεμπέκ και την Όταβα που μοιάζει να είναι προμήνυμα τέλους της παραγωγής αμύαντου. Μετά από τόσα χρόνια φαίνεται ότι η εξόριξη αμύαντου σταμάτησε στον Καναδά. Αυτό είναι θαυμάσιο ρώσιμα. Και μια μεγάλη νίκη που πρέπει, για την οποία όλοι να χαρούμε. Ήπια αρκετά ποτήρια κρασί για να το γιορτάσω. Όμως στη Ρωσία και την Κίνα συνεχίζει η παραγωγή. Και στον αναπτυσσόμενο κόσμο συνεχίζεται η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες. Και σίγουρα θα αυξηθεί η παραγωγή στη Ρωσία για να αναπληρώσει την Καναδική. Θέσατε μια ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Περίπλοκη. Πιστεύω ότι θα ήταν θαυμάσιο σχέδιο για τη νέα υποεπιτροπή αμοιάντου να ασχοληθεί με αυτό. Ξεκινώντα να εξετάσουν το θέμα αυτό, να δούνε ποιε είναι οι οικονομικέ επιπτώσει τη αφαίρεση ε, λοιπόν του αμοιάντου από όλη μα την υποδομή. Να κάνω εγώ μια ερώτηση σε εσά. Ποιο είναι το κόστο αν δεν εξηγιάνεται τα σχολεία. Πόσοι ε, δάσκαλοι και μαθητές θα πεθάνουν από απόλυτα ε, αποφεύξιμες ασθένειες. Εάν σκεφτούμε την υγεία μας, τότε πρέπει να αναλάβουμε αυτό το καθήκον, να καθαρίσουμε τα σχολεία μας, να καθαρίσουμε τα κτηριά μας, ούτως ώστε οι μελλοντικές γενιές να ζήσουν μια ζωή χωρίς αμύαντα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λοιπόν ε, ιδιαιτέρως ε, για τις παρουσιάσεις σας. Νομίζω ότι μας βοήθησαν πολύ για την έκθεση πρωτοβουλία μας. Να ρωτήσω τον εισηγητή αν θα ήθελε να πει κάτι. Ευχαριστώ τους προσκεκλημένους για τις ε, πολύ καλές ερωτήσεις, συγγνώμη, απαντήσεις στην ερώτηση θαυμάσια ιδέα να το αναλάβει η υποεπιτροπή για τον αμύαντο. Αλλά επαναλαμβάνω αυτό που είπε, είναι απαράδεκτο το κόστος του, της αδράνειας. Το θέμα είναι σε τι χρονικό ορίζοντα θέλουμε να το επιτύχουμε αυτό. Θα γίνει. Το θέμα είναι πότε θα γίνει. Εφόσον η Πολωνία έκανε την εκτίμηση και θεωρεί ότι μπορεί να το επιτύχει μέχρι το 2032, γιατί τα άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης να μην θέσουν ε, κάποιο παρόμοιο χρονοδιάγραμμα. Αλλά να το δούμε. Θα μπορούσαμε να παραγγείλουμε μία μελέτη από εξωτερικούς εμπειρογνώμενους για το κόστος και το όφελος από το καθορισμό χρονοδιαγράμματος ε, αφαίρεσης του αμοιάντου. Θα το προτείνω στην Πρόεδρό μας. Αν δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την έντονη εργασία που κάναμε. Σας εύχομαι καλή ε, επιστροφή. Αλλά πριν το κάνω αυτό, σας ρωτήσω αν υπάρχουν άλλα θέματα. Όχι, όχι. Ωραία, θα τα πούμε στις 8 ε, Οκτωβρίου για την επόμενη συνεδρίασή μας.